Eh, e Καλημέρα σε όλους και όλες. Να σας θυμίσω ότι έχουμε διερμηνία. Διαλέξτε κανάλι και έχετε. Όποια καμπίνα σας ευχαριστεί διαλέξτε. Αυτή που ανταποκρίνεται στη γλώσσα σας. Να χαιρετήσω το μεταξύ όλους σας. Τους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Καλωσορίζω για την έναρξη της συνεδριάσεως της Διακοινοβουλευτικής της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εξωτερικές Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Σας χαιρετίζω λοιπόν. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι αυτή η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια της Εβδομάδας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θέλει να την 70η επέτειο της διακήρυξης της των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η σημερινή συνάντηση θα επιτρέψει να ανταλλάξουμε εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό είναι κάτι που μπορεί να μας εμπνεύσει στις εργασίες μας ε, ως κοινοβουλευτικοί. Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που οι εθνικοί βουλευτές αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους εργασία για να καταστήσουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεσματικότερες. Πώς μπορεί όσον αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Ενώσης πιο στρατηγικές. Ποιε είναι οι ευκαιρίες, οι πιο σημαντικές, που να εφαρμοστούν για καλύτερη προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Είναι ερωτήσεις που πιστεύω ότι θα ήταν σκόπιμο να τεθούν στον προβληματισμό μας και στις εργασίες μας. Σήμερα το πρωί θα επικεντρωθούμε, θα επικεντρώσουμε το προσοχή μας σε επί τριών βασικών θεμάτων. Η πρώτη ομάδα εργασίας θα συζητήσει το πώς να εντάξουμε καλύτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εξωτερική δράση. Η δεύτερη θα επικεντρωθεί επί των βασικών προκλήσεων και τις ευκαιρίες που υπάρχουν όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, Business and Human Rights είναι το τίτλος και τρίτη ομάδα για τη βιώσιμη ανάπτυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη συνεισφορά του IYY ε, που είναι καλλιτέχνης και ακτιβιστής Κινέζος. Λοιπόν, κάποιες παρατηρήσεις θα να κάνω εδώ στην αρχή. Το στατικικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και το σχέδιο δράσεως για το 2014 μέχρι το 2019 επιβεβαιώνουν εκ νέου τη δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω να εφαρμόσει εξωτερική πολιτική που είναι πιο συνεκτική, αποτελεσματική και ορατή στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθορίζοντα στόχου και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, με ιδιαίτερη έμφαση που θα δίδεται στο θέμα της ενισχύσεως του ρόλου των τοπικών φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και ενίσχυση συνεργασίας με τους διάφορους μηχανισμούς προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο περιφερειακό και σε επίπεδο ΟΗΕ προωθώντα τα δικαιώματα των γυναικών, ένα θεματολόγιο συνεκτικό για την προώθηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων και να προωθήσει στα πλαίσια των επιχειρήσεων τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση εδραζόμενη από των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ε, πρόληψης και αποφυγής των κρίσεων και των συγκρούσεων. Κάθε κράτο μέρο θα έχει ιστορική πολιτική που θα, επι, θα επικεντρώνεται επί κάποιων πτυχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επί κάποιων συγκεκριμένων χωρών. Στην πρώτη ομάδα εργασία θα ήθελα ιδιαίτερη προσοχή να δώσουμε στην ενίσχυση και την ένταξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο κρατών μελών. Τα 28 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζουν όλη την καθολική αυτή διακήρυξη και έχουν δεσμευτεί τα κράτη-μέλη για την τήρηση αυτών των κανόνων και πρόθεση αυτών. Θα πρέπει να συζητήσουμε πώς μπορούμε να φροντίσουμε ώστε αυτέ οι αρχές να παραμείνουν προστατευμένες, εδρεωμένε και προωθούμενε στις εξωτερικέ μας δράσεις. Όπως γνωρίζετε ζούμε στιγμέ ιστορικέ, όπου οι αξίε οι αρχέ και η πολυμερής προσέγγιση αμφισβητούνται και το μέλλον των κοινωνιών μας είναι αντικείμενο μιας πολιτικής συζήτησης ζωηρής και καμιά φορά ξαναμένη συζήτησης. Όμως μπορώ να πω, πιστεύω, ότι τα δικά μας δημοκρατικά συστήματα επιτρέπουν μια συζήτηση ανοιχτή, άνευ ε, συνεπιών, ε, διαφορετικά από ό,τι γίνεται σε πολλές χώρες που δεν ανήκουν στο σίγουρο δημοκρατικό χώρο που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορούμε λοιπόν να κάνουμε βήματα συγκεκριμένα πρόοδου όσον αφορά τι προτεραιότητε που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στι εξωτερικέ μα δράσει σε επίπεδο διμερέ, πολυμερέ. Θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η αποψή σα σχετικά με αυτό. Πώ να βελτιώσουμε τι προσπάθειε που καταβάλουμε συλλογικά όσον αφορά το διεθνέ προσκήνιο και πώ τέλο μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο εθνικός και συλλογικός αντίκτυπος που παράγουμε συμβάλλει με μεγαλύτερο τρόπο ε, στην πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα να παρουσιάσω τι συνιστώσει του συμμετέχοντε στην τη Μαδαγασία. Έχουμε τον κ. Σταύρο Λαμπρινίδη, που είναι ειδικό εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον ευχαριστώ για την παρουσίαση του εδώ. Και την Πέτρα Σαστρεβίτσιου, συνάδελφο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που φέτο ήταν εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια έκθεση ετήσια όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με το Σταύρο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνιο. Ναι, χαίρομαι πολύ που σας συναντώ, αγαπητοί φίλοι. Νομίζω ότι η, ο ηγετικό ρόλο τη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι εμφανή, δεδομένη και τη παρουσία όλων ημών εδώ σήμερα για να συζητήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Πάντοτε ε, θαύμαζα τη δουλειά τη Υποεπιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και ε, βλέποντας τους πρόσφατους, ε, βραβευθέ, τους προσφάτους με το ε, βραβείο ειρήνης Νόμπελ, την Άντια Μουράτ και την Άντια Μελάλα πριν από αυτό, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το βραβείο Ζαχάροφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε δοθεί σε όλους αυτούς πριν λάβουν και το βραβείο Νόμπελ στη συνέχεια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ηγετικό ρόλο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, θα έλεγα μέσω των αντιπροσωπιών του, μέσω των ε, επιγόντων ψηφισμάτων του και κυρίως μέσω του έργου αυτής της υποεπιτροπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν που με καλέσατε σήμερα. Όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά στο εισαγωγικό σημείωμά σας, ε, ε, μπορεί να έχουμε κάποια σημαντικά σημεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά ζούμε σε έναν κόσμο όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν αντικείμενο επιθέσεων σε πολλές χώρες. Και το χαρακτηριστικό αυτή τη εποχή σε σχέση με το τι συνέβαινε πριν από λίγα χρόνια είναι ότι αυτέ οι χώρε που επιτίθεται κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι ικανοποιημένε ε, μόνο αν ζητήσουν από από ε, αυτούς που υπεραμείνονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να τους αφήσουν να ε, καταπιέζουν ε, τους πολίτες τους και να καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά προσπαθούν και να εξάγουν τις δικές τους πρακτικές σε γειτονικές χώρες, είτε σε γειτονικές χώρες άμεσα, είτε σε χώρες στις οποίες επενδύουν χρήματα, είτε σε πολυμερείς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη. Εν ολίγης, λοιπόν, θα έλεγα, Αντωνίο, ότι αυτό το οποίο έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε στην εξωτερική πολιτική ε, είναι ότι ταυτόχρονα και προσπαθούμε ε, να είμαστε ε, και διαφορετικοί χωρίς να είμαστε επιθετικοί και να είμαστε αμυντικοί ταυτόχρονα. Όταν λέω να είμαστε αμυντικοί εννοώ ε, όλες εκείνες τις περιστάσεις όπου πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτούς που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το πώς αντιμετωπίζουμε τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διάφορες χώρες. Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε ήπια διπλωματία και ισχυρά διπλωματικά μέσα με τρόπο συντονισμένο, πότε το ένα, πότε το άλλο ή και τα δύο μαζί, ούτως ώστε οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι απόπειρε ε, να αλλάξει το αφήγημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα αλλάξει. Όταν ε, λέω ότι προσπαθούμε να είμαστε ε, και επιθετικοί, εννοώ ότι με ένα πολύ στρατηγικό τρόπο προσπαθούμε να εξάγουμε τις δικές μας καλές πρακτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν ικανοποιούμεθα απλώς καταπολεμώντας αυτούς οι οποίοι υπονομεύουν το αφήγημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά προσπαθούμε να επιβάλλουμε το δικό μας ορθό αφήγημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα σας πω τι εννοώ εν συντομία. Το πρώτο το οποίο κάνουμε στην πράξη είναι ότι όλο και περισσότερο κάνουμε συνασπισμού σε ολόκληρο τον κόσμο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό το κάνουμε και δημιουργώντα μείζονε πολυμερεί και περιφερειακού οργανισμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο τη Ευρώπη, ο Οργανισμό για τη Συνεργασία στην Ευρώπη ή περιφερειακού οργανισμού στην Ασία, στην Αφρική κλπ. Και ε, επίσης ε, προσπαθούμε να κάνουμε αντίστοιχου συνασπισμού με συγκεκριμένε χώρες. Όταν μιλάμε για πολυμερείς οργανισμούς, δεν είναι τυχαία η έμφαση την οποία δίνουμε. Αυτοί που δεν ε, είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επί δεκαετίες προσπαθούν να υπονομεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η η Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων ναι. Δικαιωμάτων και οι περιφερειακέ διακήρυξει Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί για την Υλοποίηση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπω το διεθνέ Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ξεκινούν από την προσπάθεια να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτοί που είναι κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσπαθούν να υπονομεύσουν αυτού του οργανισμού. Γιατί από αυτού του οργανισμού και μηχανισμού προκύπτουν οι βασικέ δεσμεύσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με του περιφερειακού οργανισμού Έχουμε μια παρόμοια κατάσταση, κάπως διαφορετική όμως. Υπάρχει η Αφρικανική Ένωση που έχει μια πολύ αναπτυγμένη δομή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν δείτε τα κείμενά τους, αν δείτε το δικαστήριο το οποίο έχουν δημιουργήσει, η ε, διαμερικανική ε, δομή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ασιατική δομή ε, έχουν πολύ σωστές δομές. Και αν δείτε τα μέλη αυτών των οργανισμών, θα δείτε ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν είναι όλες χώρες που υπεραμείνονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλές από αυτές τις χώρες δεν είναι χώρες με εδρεωμένες πολιτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάποιες άλλες χώρες είναι πολύ κοντά στην δική μας αντίληψη περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι συμπαραστεκόμαστε σε αυτές τις χώρες. Έχουμε στοιχεί διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προσπαθούμε να εξάγουμε τη δική μας βέλτιστη πρακτική για όλα τα θέματα, για τη βία κατά των γυναικών, για τα κοινωνικο-οικονομικά δικαιώματα, για οτιδήποτε μπορεί να τους ενδιαφέρει. Ελπίζουμε ότι θα τους δώσουμε την δυνατότητα να γίνουν οι ίδιοι οι αυτών των ενιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τα προωθήσουν. Όλα αυτά είναι τμήμα μιας στρατηγικής δημιουργίας συνασπισμών. Και ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό αυτό αγαπητοί φίλοι είναι ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα σε καμία χώρα και σε καμιά περιφέρεια δεν θα εφαρμοστούν γιατί θα πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τους πει ότι έτσι πρέπει να κάνουν. Και μπορεί να έχουμε μεν και ε, μέσα πίεσης, γιατί έχουμε και οικονομική, οικονομικά μέσα πίεσης. Δεν είμαστε μία από αυτές τις δυνάμεις παγκοσμίω που χρησιμοποιούν στρατιωτικές δυνάμεις. Μπορεί να χρησιμοποιούμε ε, ενδεχομένως κάποιες κυρώσεις, αλλά όχι σε ευρία κλίμακα. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι ε, οι παγκόσμιοι και περιφερειακοί οργανισμοί που προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, μπορούν να έχουν τα μέσα να προωθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και προσπαθούμε να δημιουργούμε στρατηγικού συνασπισμού και ε, εστιάζοντα σε χώρες, όχι περιφέρειες, όχι πολυμερή συνεργασία, σε χώρε λέω τώρα, στι οποίε υπάρχει μια γκρίζα ζώνη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό παρακαλώ να το σημειώσετε σήμερα μπορεί εύκολα να μπορεί κανείς να εντοπίσει τις χώρες οι οποίες έχουν κακές πρακτικές στα ανθρώπινα δικαιώματα, χώρες οι οποίες έχουν και αναλάβει δέσμευση εναντίον των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Και εύκολα μπορείτε να εντοπίσετε και χώρες οι οποίες έχουν αναλάβει δέσμευση υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Κανείς δεν είναι τέλειος στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν δείτε όμως το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πει κανείς αυτόματα ότι αυτή είναι η κυρία κατεξοχή περιφέρεια στον κόσμο όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, είναι σε ιδιαίτερα καλή θέση. Παρατηρούμε λοιπόν αυτού οι οποίοι είναι έχουν καλέ και κακέ πρακτικέ στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά κάπω αγνοούμε τι χώρε αυτέ που βρίσκονται στο μέσο. Δηλαδή ούτε έχουν δεσμευθεί υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά μπορούν να είναι σε μια μεταβατική φάση υπέρ τη δημοκρατία χωρί να έχουν εδρεωμένες δομές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορεί να υπάρχει κάποια τάση της κυβέρνησης ε, των χωρών αυτών ε, να αντιδρά ακόμη και βία κατά ε, οργανώσεων των πολιτών οι οποίες επικρίνουν την κυβέρνηση. Μπορεί να υπάρχει επιθυμία για τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά δεν υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο δικαστικό ή άλλο. Αυτές οι χώρες στην κρίζα ζώνη είναι χώρες στις οποίες προσεγγίζουμε με μια πρωτοβουλία που είναι η πρωτοβουλία μας με τα ε, ορθά αφηγήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο φέτος ε, τα Ηνωμένα Έθνη με τον ε, πρόεδρο Αντώνιο, τον Γενικό Γραμματέα Αντώνιο Γκουτιέρε, με τη Μισελ Μπατσελέτ, είπα διαρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τη Φεντερίτα Μογκερίνη, με 13 ε, υπουργού από χώρε που συμμετείχαν από ολόκληρο τον κόσμο. Από ολόκληρο τον κόσμο, Λατινική Αμερική, Ασία, Αφρική, από την Ανατολική γειτονία, Νότια γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οκεανία. Αυτό το οποίο θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτή την ιδεολογική μάχη τη μάχη που κάνουμε εναντίον των κακών που προσπαθούν να πείσουν τους άλλους, ιδίως αυτούς που βρίσκονται σε μια ενδιάμεση κατάσταση, προσπαθούν να τους πείσουν ότι είναι κακό πράγμα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ότι σε πολλές χώρες ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν καλά παραδείγματα, καλές πρακτικές που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν πολλές κυβερνήσεις ε, που βλέπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, ως ένα στοιχείο το οποίο δεν είναι κατά της ασφάλειας, είναι ένα στοιχείο υπέρ της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, είναι υπέρ της ασφάλειας, δεν είναι εμπόδιο για την οικονομική ανάπτυξη, αντιθέτως είναι εγγενές τμήμα της οικονομικής ανάπτυξης και βλέπουν την κοινωνία των πολιτών ως ένα θεμελιώδη παίκτη ε, σε αυτό το παιχνίδι με τις κυβερνήσεις. Και στέλνουμε αυτό το μήνυμα σε όλες τις χώρες, σε ολόκληρο τον κόσμο. Χτίζουμε λοιπόν τέτοιους συνασπισμούς και θα συνεχίζουμε να εδραιώνουμε τέτοιες συνεργασίες στα επόμενα χρόνια. Το δεύτερο πράγμα που κάνουμε είναι ότι βοηθάμε την κοινωνία των πολιτών, διότι η κοινωνία των πολιτών είναι ο κατεξοχήν ιδιοκτήτης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο, εάν τα καταφέρουν να δουλέψουν σωστά σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι εδραιώνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενστερνίζονται οι πολίτε στα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό ακριβώ είναι αυτό που δεν αρέσει στι κυβερνήσει που είναι κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γι' αυτό στρέφονται και κατά ενώσεων τη κοινωνία των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κατεξοχήν υποστηρικτή τη κοινωνία των πολιτών σε ολόκληρο τον κόσμο και όχι μόνο οικονομικά, γιατί έχουμε ένα μεγάλο ταμείο που υποστηρίζει πρωτοβουλίε τη κοινωνία των πολιτών, αλλά και από πολιτική άποψη σε όλες τις επισκέψεις της ε, είπα της εκπροσώπου Φεντερίτα ε, Μοργκερίνη ή και δικές μου επισκέψεις ή και επισκέψεις όλων των ηθινόντων σε όλες τις χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο φροντίζουμε να συναντάμε σε ίση βάση εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών όπως και εκπροσώπους των κυβερνήσεων. Πολύ συχνά ξεκινάμε κοινωνικό διάλογο και έχουμε πολύ συχνά επιτύχει να φέρουμε τις ενώσεις κοινωνίας των πολιτών σε συζητήσεις με τις κυβερνήσεις. Κάτι στο οποίο αντιδρούσαν πολλές κυβερνήσεις ολόκληρο τον κόσμο, γιατί δεν ήθελαν να βλέπουν ως ίσες τις ε, ε, οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών. Τελικά όμω το αποδέχονται γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται εκεί και του λέει ότι πρέπει να το κάνουν. Προστατεύουμε του υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδίω όταν απειλούνται και παρακολουθούμε την ε, δραστηριότητά τους και δημιουργούμε μηχανισμούς προστασίας στις χώρες τους για να τους βοηθήσουμε. Νομίζω ότι ξεπέρασα ήδη το χρόνο που είχα διαθέσιμο. Θέλω κλείνοντα να πω το εξή. Εστιάζουμε στα κοινωνικο-οικονομικά δικαιώματα και στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό και είναι κομμάτι της στρατηγικής μας είναι ότι τα περισσότερα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και σχετικά με τα οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα είναι ψηφίσματα τα οποία συντάσσονται και προτείνονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ συχνά ακούγονται κριτικές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι μόνο ενδιαφέρονται για τα πολιτικά δικαιώματα και όχι για τα οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα. Δεν ισχύει αυτό και μάλιστα έχουμε διαπιστώσει ότι η αξιοπιστία μας αυξάνεται πάρα πολύ όταν εστιάζουμε σε οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα και γίνεται η αξιοπιστία μας ε, μεγαλύτερη διότι στην ε, Οικουμενική Διακήρυξη δηλώνεται σαφέστα ότι όλα τα δικαιώματα είναι αλληλένδετα. Και ακριβώς αυτό ισχύει, είναι αλληλένδετα όλα τα δικαιώματα και το θεματολόγιο για το 2030 και για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Ένωση φρόντισε τα ανθρώπινα δικαιώματα να έχουν ενσωματωθεί παντού. Και υπάρχει τώρα ένα ενιαίο κείμενο, το οποίο είναι ισχυρό, έχει γίνει αποδεκτό από όλες τις χώρες ολόκληρο τον κόσμο, εστιάζει στην ανάπτυξη στο πλαίσιο και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά είναι σπουδαία πράγματα, δεν είναι λεπτομέρειες, δεν είναι γραφειοκρατικά στοιχεία. Σε μια εποχή που οι χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο προσπαθούν να συρρυκνώσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, εμείς έχουμε κατορθώσει να επεκτείνουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τα γιγαντώσουμε. Και γι' αυτό είπα ότι είμαστε ε, σε ενεργό δράση χωρίς να είμαστε επιθετικοί. Τέλος, θέλω να πω ότι όταν επισκέπτομαι χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως επισκέπτεστε και εσείς με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακούω πολύ συχνά, όταν δεν έχουν πια άλλα επιχειρήματα να αντιπροτείνουν, μου λένε ποιος είστε εσείς κύριε Λαμπρινίδη που μας μιλάτε, ποιοι είστε εσείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση μου κάνουν την ερώτηση αυτή όταν θίγουν θέματα όπως η μετανάστευση, η ριζοσπαστικοποίηση, ο εξτρεμισμός στην Ευρώπη. δεν λένε ελάτε να λύσουμε τα προβλήματά μας, τα κοινά μας προβλήματα. Αυτό που λένε είναι ότι κάτσε στην άκρη, μην ασκείς κριτική για να μην ασκήσω κι εγώ κριτική. Εγώ όμως κάθε φορά αντιστρέφω το ερώτημα και σας παροτρύνω να κάνετε κι εσείς το ίδιο. Διότι ναι, όντως υπάρχουν προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά προσέξτε, διότι υπάρχει η παγίδα, υπάρχει ο κίνδυνος του να κάνετε ψευδείς αντιστοιχίες. Υπάρχουν κάποια στοιχεία στα οποία δεν είμαστε τέλειες και μπορείτε να πείτε «Α, και εμείς έχουμε προβλήματα, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε». Κανείς δεν είναι τέλειος, αυτό είναι αλήθεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι έχουν τις ίδιες ατέλειες στα ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα ποια είναι η λιδία λήθος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι το θέμα του αν είναι κανείς τέλειος ή όχι. Και αυτό που λέω εγώ στους συνομιλητές μου σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ότι αυτό που πρέπει να εξετάσουμε είναι θέλετε να αντιμετωπίσετε τα σημεία στα οποία δεν είστε τέλειοι ή θέλετε να τα κρύψετε κάτω από το χαλί. Θέλετε να έχετε ανεξάρτητους θεσμούς που θα σας ε, ενδυναμώνουν ε, θεσμούς που δεν θα επιτρέπουν ε, να μπαίνει κανείς στη φυλακή και να ξεχνιέται για πάντα. Έχετε ανεξάρτητα δικαστήρια, έχετε ανεξάρτητα κοινοβούλια, έχετε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, έχετε ανεξάρτητες εθνικές αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή έχετε κοινωνία των πολιτών ανεξάρτητη που μπορεί και να σας υποστηρίξει και να σας επικρίνει, να σας επικρίνει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορεί να διαφωνείτε γι' αυτό, αλλά θα τους επιτρέψετε να υπάρχουν και να σας επικρίνουν, διότι πολλές φορές σας υποχρεώνουν να γίνετε καλύτεροι. Και τελικά, αυτό είναι κάτι σημαντικό το οποίο πρέπει να τονίσουμε ότι κάνουμε. Δηλαδή, δημιουργούμε θεσμικά όργανα. Εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουμε πού υπάρχουν προβλήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και συνενώνουμε προσπάθειε με όλου αυτού που είναι πρόθυμοι να δουλέψουν μαζί μα για να δημιουργήσουμε θεσμού που θα βοηθήσουν, ούτω ώστε να μην υπάρχουν κάποιοι που δεν μπορούν να μιλήσουν. Πρέπει όλοι να μπορούν να μιλήσουν. Είναι σημαντικό να υπάρχει αρχή της λογοδοσίας και για μας και να φροντίσουμε και οι άλλοι να λογοδοτούν συνεργαζόμενοι, να βοηθήσουμε όλες τις χώρες να, να έχουν καλύτερες πρακτικές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν και αξίες τις οποίες δεν πρέπει να ξεχνάμε. Τονίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, Τονίζουμε το ότι έχουν υπογράψει τις διακηρύξεις τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να τα εφαρμόσουν και είναι, ακουγόμαστε σαν δικηγόροι γιατί πρέπει να τονίζουμε και την νομική πτυχή γιατί είναι διεθνές δίκαιο σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά δεν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα που ξεκίνησαν από το μυαλό των νομικών, ξεκίνησαν από τα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Επομένως τα ανθρώπινα δικαιώματα αντικατοπτρίζουν αξίες η ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε όλους τους πολιτισμούς και σε όλες τις θρησκείες είναι θεμελιώδες συστατικό των θρησκειών. Μπορεί στην Αφρική να το λέμε γούντου και να μην το λέμε θρησκεία. Είναι κάτι όμως το οποίο υπάρχει σε όλες τις έννοιες θρησκείας και κάθε φορά που παλεύουμε για τα δικαιώματα οποιοδήποτε ατόμου, οποιασδήποτε μειοψηφία, δικαιώματα τα οποία καταπατούνται από αυτού που δεν συμπαθούν τη μειονότητα αυτή, να θυμάστε ότι δεν υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα αυτών των συγκεκριμένων ανθρώπων και μόνο. Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα κάθε κοινωνία να δημιουργήσει ένα χώρο σεβασμού και πολυσυλλεκτικότητας και αγάπης, γιατί αυτές είναι οι κοινέ αξίες. Ο Μαντέλα είχε πει αν μπορείς να μάθεις να μισείς, γιατί κανείς δεν γεννιέται γνωρίζοντας πώς να μισεί. Αν μπορείς να μάθεις να μισείς, σίγουρα μπορείς να μάθεις και να αγαπάς. Πρέπει να διδάξουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους να αγαπάμε. Σε αυτόν τον κόσμο με τις τόσες διαιρέσεις πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε και αυτό κάνουμε βήμα-βήμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Σταύρο. Πέτρας. Ευχαριστώ Αντώνη. Αγαπητέ Σταύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπνευσμένη σου ομιλία ως προς την καθημερινή σου εργασία. Συνάδελφοι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που βρίσκεστε σήμερα μαζί για να εορτάσουμε την ε, Εβδομάδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι μια μεγάλη ημέρα. Τον τελευταίο καιρό είχαμε ε, ορισμένες ε, αντικσότητες στον τομέα αυτό. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να σας υπενθυμίσουμε πόσο σημαντικό είναι το όλο θέμα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κοινό μας αγώνα. Όπως γνωρίζετε, η συζήτησή μας εστιάζεται στην θεσμοθέτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εξωτερική δράση των κρατών μελών. Αυτό το mainstream έχει μεγάλη σημασία έτσι ώστε να ενσωματώσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον προγραμματισμό και στις επιχειρησιακές δραστηριότητες. Τη στιγμή που η θεσμοθέτηση αυτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κινείται πέρα από τη ρητορική, έχει να κάνει με μία ενιολογική βάση αλλά και με προσκόμματα όπως ανησυχίες και αμφιβολίες για το πώς μπορούμε να εντάξουμε τις, ε, το διεθνές νομοθετικό πλαίσιο στα δικά μας προγράμματα. Σήμερα προσμένω να συζητήσουμε αυτά καθώς και άλλα ζητήματα καθώς ε, και το τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι θα έπρεπε να κάνει, καθώς και τα εθνικά κοινοβούλια, έτσι ώστε να έχουμε μία καλύτερη θεσμοθέτηση των δικαιωμάτων αυτών στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει μέσω των διαθεσμικών σχέσεων έτσι ώστε και οι άλλοι οργανισμοί της Ευρώπης να λάβουν υπόψη αυτό το συσχετισμό με τις τρίτες χώρες. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ετήσια έκθεσή του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο αποτελούν ένα έγκυρο μέσο για να κατανοήσουμε κατά πόσο οι προσπάθειές μας για την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Την ε, προηγούμενη εβδομάδα στην ΑΦΕΤ εγκρίναμε την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2017. Ε, χαίρομαι που ήμουν εισηγητής και στην έκθεση αυτή η ΑΦΕΤ πρόθεσε κοινή δράση με μεγάλη πλειοψηφία των μελών που υποστήριξαν αυτό το προσχέδιο. Γι' αυτό προσμένω την έγκριση το Δεκέμβριο στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια, για να έχουμε την τελική έγκριση αυτής της έκθεσης λάβαμε υπόψη τις πραγματικές προκλήσεις στις τρίτες χώρες και προβάλαμε και προτάσεις που έχουν μεγάλη σημασία για μια καλύτερη κοινοτική ανταπόκριση. Επίσης, μιλήσαμε για την ένταξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές με εξωτερική διάσταση, όπως η ανάπτυξη, η μετανάστευση, η ασφάλεια, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, τα, ανθρώπινα, τα δικαιώματα των γυναικών και η διεύρυνση, ιδιαίτερα στον ε, τομέα του εμπορίου. Φυσικά, αυτό είναι ύψης της σημασίας για να ορίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εξωτερική πολιτική. Συνάδελφοι, τα Εθνικά Κοινοβούλια και τα κράτη-μέλη μπορούν να αντιδράσουν και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποτελέσουν υπόδειγμα προωθώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα για ολόκληρο τον κόσμο. Μόνο με την ελευθερία του λόγου και ελευθερία του συνεταιρίζεστε θεωρούμαστε ένας σημαντικός παίκτη στη διεθνή σκακέρα. Επίσης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μιλούν με μία φωνή. Θα πρέπει να έχουμε μία, έναν καλύτερο συντονισμό της εξωτερικής πολιτικής, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα στον κόσμο. Έχουμε πολύ θετικά παραδείγματα αυτής της συντονισμένης δράσης Ας δούμε την περίπτωση του, της δηλητηρίασης του Σκρίπαλ στο Σάλισμπερι του Ηνωμένου Βασιλείου, εκθέτοντας ε, τους ε, Ρώσους πράκτορες με διεθνείς κυρώσεις και από την ε, Γαλλία και τη Γερμανία. Ένας άλλος τρόπος είναι η εφαρμογή κοινών προτύπων όχι μόνο κυρώνοντας ε, διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά διασφαλίζοντας τη σωστή και έγκαιρη εφαρμογή τους. Τέτοια θέματα όπως ε, το διεθνές εμπόριο όπλων δεν αφορούν μία απόφαση ενός κράτους μέλους, διότι έχει επιπτώσει σε ολόκληρο τον κόσμο. Επιπλέον θέλω να τονίσω τη θετική, το θετικό αντίκτυπο τις ε, δράσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις σχέσεις γειτονίας. Όλα ξεκινάνε από τους ανθρώπους. Θα ενισχύσουμε το συμμετοχικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και θα προσδώσουμε τους κατάλληλους πόρους έτσι ώστε να προωθήσουμε τους υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος και πιο σημαντικό στη δράση μας είναι να αντλήσουμε διδάγματα από τα, την πρακτική αυτή ως προς την εξωτερική πολιτική διεύρυνση και πολιτικές γειτονίας για να προωθήσουμε τις διαθεσμικές σχέσεις και διακοινοβουλευτικές σχέσεις που είναι ύψης σημασίας. Κυρίες και κύριοι, χωρίς να καθυστερούμε, θα ήθελα να προχωρήσουμε στη συζήτηση την οποία προσμένω και εγώ και είμαι σίγουρος ότι η ανταλλαγή απόψεων θα αποτελέσει μια κοινή βάση αξιών για τη συνεργασία μας επί του θέματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πέτρα. Έχουμε μισή ωρίτσα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε στα πλαίσια του πρώτου πάνελ. Γι' αυτό θα παρακαλούσα τους συναδέλφους που θέλουν να παρέμβουν να μην ξεπεράσουν τα δύο λεπτά ο καθένας, όπως έχουμε συνηθίσει στο Κοινοβούλιο, ούτως ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα να δοθούν και κάποιες απαντήσεις από πλευρά των φιλοξενουμένων μας. Πρώτος που θα πάρει το λόγο, ο συνάδελφος Μόρεν από την Ιρλανδία. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μπορέσω να μιλήσω εδώ. Καταρχάς πρέπει να δεχτούμε το ρόλο που έξε η Ιρλανδία με, στις διαπραγματεύσεις την Κένια για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της Κένιας για να εξασφαλίσουν συμφωνία και τη διαπραγμάτευση των στόχων ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Να πω και κάτι για την Ιρλανδία ότι η βοήθειά μας εστιάζεται επί της φτώχειας. 100% ε, είναι αδέσμευτη. Δεν ζητάμε κάτι σαν αντάλλαγμα και συνεργαζόμαστε με τι πιο φτωχέ και ευάλωτε χώρε στον κόσμο. Και νομίζω είμαστε σε μοναδική θέση λόγω τη ιστορία μα να το κάνουμε αυτό. Ποτέ δεν ήμασταν απικιακή χώρα. Εμεί ε, δεχτήκαμε απεικιοκρατία και ήμασταν θύματα τη πείνα και μαζική ε, αποδημία των κατοίκων. Λοιπόν, οι λέξει θα πρέπει, που είναι ιδεολογικά φορτισμένε και σωστά φορτισμένε πρέπει να ακολουθηθούν από πράξη. Κάποιοι τομεί βλέπουμε μεγάλε αντιφάσει από χώρε που μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα. Και να αναφέρω κανένα δύο παραδείγματα. Πρώτα απ' όλα είναι το εμπόριο περιόπλων. Οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και χώρε του ΟΗΕ που τροφοδοτούν το εμπόριο όπλων, το οποίο συμβάλλει στην αύξηση τη στόχια, τη πείνα και του εκτοπισμού. Ε, η έλλειψη πραγματικής ε, δικαιοσύνης φορολογικής χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΟΗΕ, που διευκολύνουν το ότι ο Νότος ε, χάνει πολλά χρήματα κάθε χρόνο. Η άλλη αντίφαση αφορά την αλλαγή του κλίματος Ακόμα δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν πάνω σε αυτό όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος. Και βλέποντας την αυξανόμενο το θεματολόγιο που εξετάζει περισσότερο την ασφάλεια, ο στρατός δεν συμβάλλει στη μείωση της φτώχεια και της πείνας και των συγκρούσεων. Προσθέτουν σε αυτά τα φαινόμενα, αλλά βλέπουμε τώρα αυξανόμενο θεματολόγιο ενισχύσεως της ασφαλείας. Το είδαμε αυτό το παράδειγμα στη Μεσόγειο και πρέπει να ρωτήσω, πού είναι το θεματολόγιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν κοιτάμε προς την Μεσόγειο. Είμαστε πολύ καλά στο να λέμε λόγια, λόγια, λόγια, αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε τα λόγια πράξη. Και δεν θα πρέπει να είμαστε αντιφατικοί στι πολιτικέ μα. Δηλαδή να δίνουμε το ένα χέρι και αυτά που δίνουμε τα παίρνουμε το άλλο χέρι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλο συνεισφορέα όσον αφορά τη χορήγηση βοήθεια, αλλά συμβάλλουμε και στα εργοστάσια που είναι τα αίτια τη ανάγκη για βοήθεια. Πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα εμεί τι κάνουμε. Διότι κανεί τελικά δεν μπορεί να πει ότι είναι τέλειο. Νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε πάρα πολύ καλύτερα. Δηλαδή, ε, ε, αυτό κάνουμε, δηλαδή είμαστε δίγλωση. Ε, και αυτή η δίγλωση πρέπει να σταματήσει. Συνάδελφε Σούσκιν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ, όπως και η συνάδελφός μου την Ιρλανδία, και εγώ θέλω να συμφωνήσω με αυτά που είπε και τα θέματα που έθεσε. Θα ήθελα να τονίσω εδώ την κατάσταση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέποντας την αύξηση των αντιφιλελεύθερων τάσεων, αντιδημοκρατικών τάσεων σε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό προφανώς δυσχεραίνει κατά πολύ ε, την τοποθέτησή μας στην εξωτερική πολιτική. Ερώτηση, πώς βλέπετε αυτές τις πολύ ανησυχητικέ εξελίξεις, διότι μπορούμε να κάνουμε παραλληλισμούς μεταξύ αυτών που συμβαίνουν στη Ρωσία, με αυτά που συμβαίνουν εντός αρκετών χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σε άλλες χώρες, όπως είπε και συνάδελφο, Μπορούμε να μιλήσουμε την Αίγυπτο και το Ισραήλ, που είναι μια δημοκρατία που εφαρμόζει όμω πολιτικέ που θέτουν εν κινδύνο το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή η κατάσταση ήταν ε, πολύ ε, λιγότερο ε, στεναρή τα προηγούμενα έτη. Έχει σχηροποιηθεί τώρα. Θέλω να ξέρω ποια είναι η άποψή σα γι' αυτό. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Πρέντα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να χαιρετήσω την παρουσία του πρώην συναδέλφου μας, του Σταύρου Λαμπρινίδη εδώ. Δύο λόγια θέλω να πω όσον αφορά το ερώτημα που ετέθη μόλις τώρα για να αναφέρω κάποια εργαλεία που το Κοινοβούλιο μας ε, χρησιμοποιεί για να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καταρχάς έχουμε την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που υθετούμε προς το τέλος κάθε χρόνου και πρέπει να πω ότι την ε, πρόσφατη περίοδο όλο και περισσότερο τονίσαμε το θέμα της δημοκρατίας. Ξεκινώ την ιδέα ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για το σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτός του δημοκρατικού πλαισίου. Ε, βλέπουμε συμπεριλαμβανομένε και τι εκθέσει που ετοιμάστηκε από το φίλο Στροβίτσιου, που ετοιμάστηκε φέτο, βλέπουμε αυτή τη σχέση που υπάρχει και υπογραμμίζεται. Δεύτερον, να επενθυμίσω και κάτι άλλο, ότι κάθε μήνα υιοθετούμε ψηφίσματα στα κατεπήγοντα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύω ότι αυτό είναι μοναδικό στην Ευρώπη. Ε, δεν περνάνε αυτά σε επίπεδο εθνικό. Θα ήταν ενδιαφέρον να ανταλλάξουν πόψει με του βουλευτέ που έρχονται από τα εθνικά κοινοβούλια. Γιατί δεν γίνεται αυτό σε εθνικό επίπεδο. Στο Στρασβούργο κάθε μήνα ετοιμάζουμε ψηφίσματα στα κατεπήγοντα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι παρόμοιο σε επίπεδο των εθνικών κοινοβουλίων. Τρίτον, θα ήθελα να αναφέρω τις διάφορες ακροάσεις που διοργανώνουμε εδώ ή στο Στρασβούργο πάνω στα θέματα των ε, δικαιωμάτων. Πώς να το πω. Σε κάποια εθνικά κοινοβούλια γίνεται το αντίστοιχο. Γίνονται ακροάσεις, hearings όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά δεν γίνεται παντού αν δούμε τι γίνεται σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Να επενθυμίσω ότι κάθε χρόνο Δίνουμε το, απονέμουμε το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης και φέτος θα δώσουμε αυτό το βραβείο στον Όλεξ Ένσοφ, έναν Ουκρανό σκηνοθέτη που ξέρει όλος ο κόσμος. Να πω τέλος ότι κάθε χρόνο ασκεί δραστηριότητες εποπτείας εκλογών, παρατηρήσεις εκλογών. Και αυτό τίθεται πάντα στα πλαίσια του σεβασμού των δικαιωμάτων. Σε αυτό το επίπεδο Υπάρχει μία συνεργασία με τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων μέσω των διαφόρων μορφών, σχημάτων και κυρίως με τους βουλευτές που προέρχονται από τα κράτη-μέλη στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ΟΑΣΕ. Αποστολές επιτηρήσεως των εκλογών, ελέγχου των εκλογών. Αυτά είναι κάποια εργαλεία που διαθέτουμε και θα ήμουν ενδιαφέρον θα είχε ενδιαφέρον να αλλάξουμε απόψει με του συναδέλφου, να δούμε πώ να συγχρονίσουμε τι δράσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τι δράσει στα διάφορα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφε Πέτα. Συνάδελφε Κάν, έχετε το λόγο. Uh, thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ξανά το Σταύρο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνεις και για όλες τις προσπάθειες που καταβάλεις ως ειδικό εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συμφωνώ με αυτά που είπες και θα επαναλάβω αυτό που είπες και εσύ για το Μαντέλα. Ο Μαντέλα ε, ποτέ δεν έχασε την ελπίδα. και τόνισε αυτή την εικόνα που είχε δώσει και ο Βρετανός ε, Φρέντερικ Βότς. Είναι πραγματικές οι ανησυχίες για το μέλλον, βλέποντας την κατάσταση του κόσμου μας σήμερα. Στο πλαίσιο των εξωτερικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι ότι αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε σχέσεις φιλίας και συνεργασίας. Το θεματολόγιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πώς θα το κρατήσουμε σε υψηλή θέση στις προτεραιότητές μας. Αν πάρουμε την Κίνα και την Ινδία, δύο μεγάλες αναδυόμενες δυνάμεις, βλέπουμε το τι γίνεται στην Κίνα, εδώ, στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έρχονται άνθρωποι που μας παρουσιάζουν ε, περιπτώσεις καταπίεσης ε, και ε, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και στις περιοχές της Ινδίας, όπως το Κασμίρ, δεν επιτρέπεται πολύ συχνά στους επισκέπτες να επισκεφθούν καν το Κασμίρ. Μιλάμε για ιστορικές διενέξεις. Μερικές φορές μπορεί να είναι και εδαφικές, όπως στην περίπτωση του Κασμίρ. Υπάρχει το θέμα της ειρήνης μεταξύ των χωρών και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα μπορούσε να είναι κομμάτι αυτής της μακροπρόθεσμης λύσης για την ειρήνευση αυτών των ε, εδαφικών διενέξεων. Δηλαδή να το συνδέσουμε αυτό με ορισμένα από τα ψηφίσματα για τα κατεπήγοντα να επιδιώξουμε και μακροπρόθεσμη επίλυση των διενέξεων και να διασφαλίσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται σεβαστά. Ευχαριστώ πολύ, Μπάρμπορα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για όλους για τις παρουσιάσεις. Έχω τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, για τα κείμενα τα οποία έχουμε που βασίζονται στους γενικούς κανόνες. Από τον, ε, έχουμε τον κύριο Μπόλτον που είναι κατά της ύπραξης του διεθνούς δικαίου και άλλες κυβερνήσεις επίσης θεωρούν ότι όταν εκπροσωπούν το λαό τους είναι πάνω από τον νόμο και δεν χρειάζεται να λογοδοτούν. Είναι δύσκολο λοιπόν το καθήκον μας και εμείς και εσείς τα Ηνωμένα Έθνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα ψηφίσματά μας και στην έκθεση που, του κ. Στρεβίτσιους, θεωρούμε ότι προσθέτοντας στη δική σας θέση που εστιάζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει και ένας ειδικό εισηγητής για την ενίσχυση του διεθνούς ε, ανθρωπιστικού δικαίου και του ε, διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί πρέπει να είμαστε περισσότερο ενεργοί και χρειάζεται μεγαλύτερη υποστήριξη σε διεθνές επίπεδο. Ελπίζουμε στην ετήσια αυτή έκθεση ε, να μπορέσει να υπάρξει μια τέτοια ε, μνήα και ελπίζω να το υποστηρίξει η Φεντερίκα Μογκερίνη. Δεύτερον, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι και στα Ηνωμένα Έθνη ε, δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε με μία και μόνη φωνή και γι' αυτό και αποδυναμωνόμαστε ως περιφέρεια. Και όπως και για το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, κράτη-μέλη αγνοούν γεγονότα. Η Αυστρία, η Πολωνία, η Ουγγαρία αποσύρονται, λένε ότι δεν θα το υπογράψουν. Λένε ότι είναι νέο δίκαιο, αλλά αυτό δεν ισχύει, απλώς συγκεντρώνουμε υφιστάμενες πολιτικές. Αποδυναμώνουμε λοιπόν την ε, επιρροή της περιφέρειάς μας με την τακτική αυτή που ακολουθούν πολλές χώρες. Και τρίτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ισχυρή περιφέρεια και λόγω της οικονομικής της επιρροής. Αυτό δεν είναι κακό, αλλά θα έπρεπε να ενισχύσουμε τη σχέση μεταξύ των εμπορικών προτιμήσεων, παραδείγματος χάρη, και της αιρεσιμότητας ε, για την βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό θα ήταν μία λύση, αντί να μιλάμε μόνο για το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν περιπτώσεις όπως η Μιανμάρ, το Βιετνάμ, η Καμπότζη και ελπίζουμε ότι η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα δείξουν κάποια αυστηρότητα για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γένσεν. Η κυρία Γένσεν. Η κυρία Γένσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση αυτή και χαίρομαι που γίνεται αυτή η συζήτηση παράλληλα, για, με, με την εξωτερική δράση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε ε, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο ένα πρόγραμμα για την ε, προστασία των κοινοβουλίων. Οι βουλευτέ προστατεύουν του βουλευτέ για να μπορέσουμε να προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάθε βουλευτή έχει την ευκαιρία να υιοθετήσει μια μεμονωμένη περίπτωση και να υποστηρίξει μια συγκεκριμένη υπόθεση για την απελευθέρωση κάποιου από μια φυλακή ή για τη δυνατότητα ενίσχυση ε, αντικαθεστωτικών. Ήθελα απλώς να αναφέρω το πρόγραμμα αυτό νομίζω ότι είναι μοναδικό σε ολόκληρο τον κόσμο και ίσως να υπάρχει και η δυνατότητα να εφαρμόσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα και άλλα εθνικά κοινοβούλια. Όχι μόνο για να τονίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε γενικό επίπεδο, τα οποία ακολουθούμε με βάση τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με μονομένες περιπτώσεις, δηλαδή να υπάρχει ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη εικόνα την οποία προωθούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Elnök úr, tisztelt... αξιότιμη κυρία Λαμπρινίδη, σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας και ως ε, πρώην συνάδελφό μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, ε, σας καλωσορίζουμε και εσά και τους βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια, τους συναδέλφους από τα Κοινοβούλια της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας. Έχω τις εξή ερωτήσεις. Πρώτον, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η προστασία τους η προστασία τους και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός. Γιατί πολύ συχνά βρισκόμαστε σε μια σχιζοφρενική κατάσταση που υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των Ουιγούρων ή του Θιβέτ, ενώ υπάρχουν πολλά ευρωπαϊκά κράτη-μέλη όπου παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα κατάφορα. Στη Ρουμανία, παραδείγματος χάρη. Ε, εγώ είμαι Ούγγρος ρουμανικής καταγωγής. Καλό θα ήταν στις δραστηριότητες της Επιτροπής και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων να τις έχουμε κατά νου ούτως ώστε να προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα δεύτερο ερώτημα τώρα, οικονομικό. Δυστυχώς έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τα οικονομικά συμφέροντα εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραδείγματο χάρη στις σχέσεις με την Κίνα. Για παράδειγμα, οι Ουιγούροι υποφέρουν και σε πολλά σημεία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι τα οικονομικά συμφέροντα παίζουν σημαντικό ρόλο και δεν έχουμε την απαιτούμενη ε, συνέπεια όταν μιλάμε για τα δικαιώματα των Ουιγούρων, του Θιβέτ ή άλλων ε, πληθυσμών σε τρίτες χώρες. Και το τρίτο μου ερώτημα που έχει σχέση με τη μετανάστευση. Το Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τη Μετανάστευση το εξετάζουμε από την πλευρά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σήμερα. Δικαίωμα στη μετανάστευση, είναι ε, ένα ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά είναι ένα είδος σκληροπυρηνισμού στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα θέματα ασφάλειας. Βεβαίως και πρέπει να αποδεχόμεθα ανθρώπους που καταφεύγουν σε εμά και να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά υπάρχουν και οικονομικοί μετανάστες. Εδώ δεν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή να μην κατασκευάζουμε ανθρώπινα δικαιώματα. διεξάγονται πολλές συζητήσεις για το Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τη μετανάστευση και εδώ θα πρέπει πολύ ανοιχτά να μιλήσουμε. Να μην ε, ε, βάλουμε κάποια θέματα ταμπού και να μην μιλάμε με δύο μέτρα και σταθμά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Συνάδελφε όλοι έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα. Όπως και κάποιοι συνάδελφοι ήδη ανέφεραν και εγώ θέλω να τονίσω κάτι. Υπάρχει ασυνέπεια μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι κάτι που μας αποδυναμώνει σχετικά με την προστασία και πρόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Συμφωνώ με τον κύριο Λαμπρινίδη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιθανότατα είναι ο τόπος όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύονται περισσότερο όμως έχουμε και κάποια ελαττώματα και κενά και προβλήματα. Αν δεν τα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, αυτό μειώνει την αξιοπιστία μας όσον αφορά τις δραστηριότητες μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάποιοι συνάδελφοι παρέθεσαν άλλα παραδείγματα. Εγώ είμαι από την Καταλωνία. Θα μπορούσα επί να αναφερθώ για τα τεκτενόμενα στη χώρα μου. Όσον αφορά τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα, Σήμερα 400 μέρες έχουν περάσει που ο Τζόρντι Κοσάρτ και ο Τζόντι Σάντσες, δύο ακτιβιστές, πολιτικοί και κοινωνικοί ακτιβιστές, μπήκαν στη φυλακή. Είναι φυλακισμένοι 400 μέρες χωρίς δίκη. Δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα ξεκινήσει η δίκη. Κατηγορούνται για επανάσταση, για στάση, διότι οργάνωσαν ε, οι ειρηνικέ διαδηλώσει, μαζικέ αλλά ειρηνικέ διαδηλώσει υπέρ τη ανεξαρτησία τη Καταλωνία. Άρα έχουμε κάποια προβλήματα εδώ, εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να τα λύσουμε αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι στα μάτια του κόσμου. Εδώ στο Κοινοβούλιο στηρίζαμε ένθερμα την ανάγκη ύπαρξης μηχανισμού, μέσω του οποίου σταθερά παρακολουθούμε την εφαρμογή των πολιτικών δικαιωμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την περασμένη εβδομάδα στο Στασβούργο εγκρίναμε ένα ψήφισμα. Σε αυτό συστήνουμε ένα τέτοιο μηχανισμό. Αν μπορούσε να υπάρξει αυτός ο μηχανισμός και υπάρχει συνεχής εποπτεία κάθε κράτους μέλους για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τότε θα μπορούσε να διευκολύνει αυτό τις δράσεις μας και τα καθήκοντά μας όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Καλώς, λέει ο Πρόεδρος. Έχετε 4-5 λεπτά ο καθένας να απαντήσετε. Ο Πέτρας πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για τη γνωμοδότησή σας και τα ερωτήματά σας. Ξεκινώντας από την Ιρλανδή εκπρόσωπο, εκτιμώ την Ιρλανδική αναπτυξιακή πολιτική προς πολλές χώρες και νομίζω ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την αναπτυξιακή πολιτική και την αποτελεσματικότητά της για να φτάσουμε στους απότερους στόχους και για να υπάρχει αυτάρκεια αυτών των χωρών που πρέπει να αναπτύξουν τη δική τους πολιτική. Θα πρέπει να συνεχίσουμε με αυτή την πολιτική για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά πάσα πιθανότητα, αλλά οι χώρες αυτές θα πρέπει να γίνουν αυτάρκειες. Συμφωνώ με αυτά που είπατε για την κατάσταση της ασφάλειας αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Η ασφάλεια βρίσκεται στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Ε, υπάρχουν ε, ε και στην Ευρώπη για πολλές δεκαετίες δεν υπήρχαν, τώρα όμως επανέκυψαν. Και δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε. Υπάρχει θέμα εθνικής και εδαφικής κυριαρχίας. Πολλές φορές οι ε, ηγέτες ε, δακτυλοδεικτούν τις γείτονες χώρες. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα σύνορα, αλλά οι άνθρωποι. Πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε αυτά τα μήνυματα και να καταλάβουμε ότι χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχει εμπόριο. Δεν υπάρχει συνεργασία. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να βασιστούμε στις διεθνείς συμφωνίες έτσι ώστε εκεί που υπάρχει παραβίαση να επανέλθουμε στην ε, τάξη. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό σύντομα. Ως προς το ερώτημα για ορισμένες ανησυχητικές εξελίξεις για πολύ καιρό οι προδιαγραφές ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν μια καθολική αξία. Αυτό που βλέπουμε όμως αυτή τη στιγμή είναι μια προσπάθεια να οριστούν εθνικές ή περιφερειακές προδιαγραφές ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ορισμένου ηγέτες που προσπαθούν να επιτεθούν στα ανθρώπινα δικαιώματα λέγοντας «Α, εμείς ε, εξαιρούμαστε». Για μας ισχύει κάτι άλλο. Τα ε, δικαιώματα των ομοφιλοφίλων δεν μας αφορούν, τα δικαιώματα των ε, γυναικών δεν μας αφορούν, η διακίνηση ιδεών δεν μας αφορά και ούτω καθεξής. Εάν κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, δεν μπορούμε να δεχτούμε τις εθνικές ή περιφερειακές αυτές προδιαγραφές. Θα πρέπει να μας απασχολούν οι καθολικές αξίες και φυσικά η περίπτωση της Ρωσίας είναι κάτι το εξειδικευμένο. Δεν μπορώ να δεχτώ τη ρωσική αυτή ιδεολογία η οποία εξάγεται ε, προς τα έξω, ιδιαίτερα ως προς την ε, πολιτική της γειτονίας. Θα πρέπει η Ρωσία να βασιστεί στις διεθνείς προδιαγραφές και να τηρήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ως προς την αιρεσιμότητα θα ήθελα να πω ότι είναι μια βασική έννοια, αλλά οι εμπορικές ε, πολιτικές και οι οικονομικές ε, προς τις τρίτες χώρες θα πρέπει να συνδεθούν με τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι ώστε αυτό να αποτελεί, αυτά να αποτελούν απαράβατο όρο ως προς την αποτελεσματικότητα της πολιτικής. Πρόσφατα, στην περίπτωση της Καμπότζης, είδαμε ότι ήμασταν πολύ εφεκτικοί και σιωπήσαμε για χρόνια. Αρνούμενοι να δούμε τα αρνητικά ε, θέματα και αποτελέσματα στην Καμπότζη. Τη στιγμή που δεν υπάρχει ελευθεροτυπία και ελεύθερα μήμη τότε μόνο προβαίνουμε σε κυρώσεις. Αυτό θα πρέπει να έχει γίνει προγενέστερα και είναι ύψης της σημασίας η έγκαιρη επέμβαση. Και θα ήθελα να πω ως προς τη Μολδαβία ε, πήραμε αρνητικά μέτρα, δηλαδή παγώσαμε τα 100 εκατομμύρια ευρώ μακροοικονομικής βοήθειας, γιατί είδαμε να μην τηρούνται οι δημοκρατικές διαδικασίες. Νομίζω ότι φυσικά ήταν μια αρνητική απόφαση, αλλά έπρεπε να ληφθεί για να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βασίζεται μόνο στο εμπόριο, αλλά στις αξίες και τη στιγμή που βασιζόμαστε στις αξίες αποτελούμε μία ήπια οικονομική δύναμη παγκοσμίω. Θα ήθελα να τονίσω και το παράδειγμα της Γερμανίας, την κοινοβουλευτική πρωτοβουλία που ελήφθη. Πολλές φορές σώζει ζωές και προωθεί τη δημοκρατία σε ορισμένες χώρες. Δηλαδή θα πρέπει να συμμεριζόμαστε αυτή την εμπειρία πριν από τη συνάντησή μας για να ξέρουμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές κάθε φορά που συναντιόμαστε και φυσικά ε, αναμένω τη μελλοντική μας συνεργασία γιατί ενέχει μεγάλη αξία. Ευχαριστούμε πολύ ο Σταύρος. Ευχαριστώ Αντώνιο. σημείωσα ότι πολλές ερωτήσεις τρέφονται γύρω από την εσωτερική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κατανοώ αυτό, γιατί όλοι μιλάτε για τη σύνδεση μεταξύ της αξιοπιστίας μας ε, και της ικανότητάς μας ε, να μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχετε δίκιο, υπάρχει αυτή η σύνδεση. Δεν είναι το κέριο το αντικείμενο αυτής της συνεδρίασης. Ε, ούτε και η δική μου εντολή το να ασχολούμαι με τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα ήθελα ε, να επαναλάβω κάποια σημεία που θεωρώ σημαντικά. Έχετε δίκιο ότι όντως αντιμετωπίζουμε προκλήσεις και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του κόσμου τον οποίο επί δεκαετίες θεωρούσαμε δημοκρατικό είναι σημαντικές προκλήσεις και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Δεν τις ε, παραβλέπω κατά κανένα τρόπο, αλλά σας διαβεβαιώ από τα ταξίδια μου σε ολόκληρο τον κόσμο όταν βλέπω παραβιάσεις ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι σοβαρές αυτές οι παραβιάσεις. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτές τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε στις δημοκρατικές χώρες που μας σοκάρουν, διότι είναι ε, εναντίον των βασικών αρχών τις οποίες συνστερνιζόμαστε. Αλλά σε άλλες χώρες θα ήταν ε, αστείες αυτές οι προκλήσεις, αν τις συγκρίνουμε με τα εγκλήματα, με τους βασανισμούς, με τους εγκλισμούς χωρίς καμία αντίδραση τηλεόραση, των μέσων ενημέρωσης ε, ή του διαδικτύου. Σας παρακαλώ λοιπόν, ε, όπως είπα και στην αρχή, να αποφύγουμε την παγίδα της ψευδούς αντιστοίχησης. Επανέρχομαι σε αυτό που σας είπα, γιατί το κάνω συνεχώς στη δουλειά μου, οφείλω να το κάνω. Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τεράστια σημασία. Και το να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι προκλήσει είναι εξίσου σημαντικό όπω και το να προασπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά α έχουμε παράλληλα κατά νου ότι ενώ αντιμετωπίζουμε τις εσωτερικές μας προκλήσεις, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να πέσουμε σε μια δεύτερη παγίδα, δηλαδή να αποθαρρυνόμεθα για τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα. Μερικές φορές όταν μιλάμε για τα εσωτερικά μας προβλήματα, σχεδόν προβάλλουμε προς τα έξω μία απόγνωση. Φαίνεται ότι δεν λειτουργεί τίποτα, ούτε στην Ισπανία, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην ε, Ουγγαρία, στην Πολωνία. Α, κοίτα τι γίνεται στην Ολλανδία, τίποτα δεν λειτουργεί. Να τα συλλητεύσουμε μένα, αλλά το αποτέλεσμα να μην είναι ότι θα νιώθουμε ότι δεν έχουμε δικαίωμα να ασχολούμεθα με τις παραβιάσεις άλλων, γιατί κοίτα τι κάνουμε εμείς. Έτσι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα παντού. Αυτοί που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρο τον κόσμο, αυτό προσπαθούν να κάνουν. Ακριβώ αυτό προσπαθούν να μα διαιρούν σε όλα τα θέματα καθημερινά. Και μέσω ψευδών ειδήσεων και μέσω πολλών μέσων θέλουν να μα στρέψουν τον ένα εναντίον του άλλου, να μα κάνουν να νιώθουμε σε απόγνωση, να θεωρούμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν προσφέρουν τίποτα, και αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, στα Ηνωμένα Έθνη είναι να πούμε ότι ε, κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά όταν το Περού μείωσε το επίπεδο φτώχειας από 55% σε 22% σε 7 χρόνια μόνο και αυτό το έκανε μέσω της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών, της κυβέρνησης ε, των ενώσεων εργαζομένων, εξασφαλίζοντας την ισότητα στην κατανομή του πλούτου, αυτό είναι ένα παράδειγμα για να το προτείνουμε να το ακολουθήσουν και άλλοι. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με το παράδειγμα της Κίνας που παραβιάζει ανθρωπίνα δικαιώματα ενώ ακολουθεί ε, πολιτική οικονομικής ανάπτυξης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν, είναι θεμελιώδη σημασία να μην πέφτουμε σε τέτοιες παγίδες. Τώρα, στο ίδιο πλαίσιο, Όντως έχουμε ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ορισμένες φορές φαίνεται ότι αντικατοπτρίζουν κάποιος ανέφερε τη Ρωσία όμως υπάρχει μια διαφορά Αυτό το οποίο βλέπω στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια είναι μια συστηματική καταπίεση κάθε φωνής που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και καταγγέλει τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων καθημερινά μπορούν να καταγγέλουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα υπάρχει διαδικασία, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές συνθήκες, ε, να ξεκινούν διαδικασίες κατά των χωρών που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στη Ρωσία ή σε άλλες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οπότε σας απαντώ ότι ναι, βεβαίως και με ανησυχούν οι παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να μην πέφτουμε σε αυτή την ε, παγίδα. Ένα δεύτερο θέμα τώρα για την ανάπτυξη και το εμπόριο. Αναφέρθηκε το σύστημα των γενικευμένων προτιμήσεων ε, ε, ΣΥΝ. Τι ακριβώς είναι αυτό το GSP+. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι λέμε σε όλες τις χώρες, σε ολόκληρο τον κόσμο, ότι θα σας αφήσουμε τα προϊόντα να έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μηδενικούς δασμούς σχεδόν, αλλά υπό έναν όρο. Και ποιος είναι αυτός ο όρος ότι οι Ευρωπαίοι απαιτούν να εξάγουν τα πορτοκάλια με μηδενικούς δασμούς κατά τον ίδιο τρόπο, ότι θα έρθουν οι μεγάλες ευρωπαϊκές κατασκευαστικές εταιρείες να κατακλείσουν τη χώρα. Ποιος είναι ο όρος αυτών των κοινικών Ευρωπαίων για να έχουμε μηδενικούς δασμούς. Αυτό μας ρωτάνε. Η απάντηση ποια είναι. Ο μόνος όρος είναι ότι πρέπει να εφαρμόζεται όλες τις διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή είναι η μοναδική συνθήκη, ο μοναδικός όρος για το GSP+. Οι χώρες αυτές λοιπόν που θα έχουν αυτές τις ειδικές γενικευμένες προτιμήσεις θα πρέπει να εφαρμόζουν και να επαληθεύεται ότι εφαρμόζουν η οικουμενική διακήρυξη, οι συνθήκες του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και όλες οι συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μοναδική περιφέρεια σε ολόκληρο τον κόσμο που βάζει στο κέντρο των εμπορικών πρακτικών της ε, τέτοιου όρου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν είναι εύκολο, σας διαβεβαιώ, γιατί σε αυτό τον ίδιο κόσμο υπάρχουν όλο και περισσότερες χώρες που έχουν χρήματα και που ευχαρίστως ε, θα χρησιμοποιήσουν και πρακτικές διαφθοράς προς ξένες κυβερνήσεις για να αποκτήσουν οικονομικά συμφέροντα. Δεν είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να ασκήσουμε οικονομική πίεση πίεση. Εμείς ασκούμε θετική οικονομική πίεση. Υπάρχουν άλλες μεγάλες δυνάμεις που ασκούν αρνητική οικονομική πίεση. Και πάντοτε πρέπει να εξετάζουμε πώς μπορούμε να εφαρμόζουμε τις υποχρεώσεις μας. Κάθε μέρα το προσπαθώ αυτό. Προσπαθώ να εφαρμόζουμε τις οικονομικές μας πιέσεις θετικά, χωρίς να χάνουμε όλες αυτές τις χώρες που ακούν τις σιρήνες των αυτών που προσπαθούν να τους προσελκύσουν με αρνητικά μηνύματα. Εμείς προσπαθούμε να εφαρμόζουμε όλη αυτή την πολιτική με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τρίτο θέμα, ασφάλεια. Ναι και μακροπρόθεσμη ειρήνη ε, θέλουμε ε, που δεν είναι σε διένεξη με τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, σε βραχυπρόθεσμο μη προοπτική. Μπορεί να φαίνονται αντιφατικά, αλλά δεν είναι. Προσπαθούμε με την πολιτική μας να προβλέπουμε τις ε, διενέξεις για να τις ε, αποφεύγουμε. Και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα από τα σημεία τα οποία εξετάζουμε για την αποφυγή των διενέξεων. Όταν υπάρχουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αντιμετωπίζονται και λαμβάνονται πάντοτε υπόψη ε, όταν ε, προσπαθούμε να επιλύσουμε κάποια διένεξη. Δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι χωριστά από την ειρηνευτική διαδικασία. Είναι στον πυρήνα της ειρηνευτικής διαδικασίας και αυτό είναι μέσα στην καθημερινή μας δουλειά. Κάποιο ανέφερε και την έννοια φορολογική δικαιοσύνη. Βεβαίω και έχετε δίκιο. Οι ανισότητες και οι οικονομικές και οι κοινωνικές παράλληλα με, τις, ε, τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα και τις αντίστοιχες ε, ανισότητες έχουν θεμελιώδη σημασία. Ε, καθημερινά βλέπουμε αυτούς που εμφανίζονται ως επιτυχημένοι ενώ αυτοί που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν την αντίστοιχη ε, σημασία. Φαίνεται να μην ενδιαφέρονται όλοι για το κοινό καλό. Πρέπει τη μάχη αυτή να την κερδίσουμε, να ενδιαφερόμεθα για τα δικαιώματα όλων ε, των ομάδων. Αυτή την αξιοπιστία που μας προσφέρει η άμυνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κάτι που παρολίγο να το χάσουμε αλλά το ξανακερδίζουμε με καθημερινούς αγώνες. Αντώνιο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά που έχεις κάνει. Ε, με θαυμαστό τρόπο διεξάγεις τις επαφές με όλα τα θεσμικά όργανα και η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακούγεται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην, εξωτερική υπηρεσία, στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Προς τον θέλω να πω ότι ε, η δουλειά την οποία έχετε κάνει ε, και φέτος ε, για να ληφθούν υπόψη όλες οι συμβαστικές λύσεις ε, πριν φτάσει στην Ολομέλεια η έκθεση, ούτως ώστε να ακουστεί η φωνή του Κοινοβουλίου ως μία ενιαία φωνή, είναι πολύ σημαντικές προσπάθειες αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μιλάει με μία και μόνη φωνή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν πρέπει να δίνουμε την εντύπωση ότι μιλάμε με χωριστές φωνές. Και το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι θεμελιώδους σημασία. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ και εσείς από τα Εθνικά Κοινοβούλια ελπίζω αυτό το μήνυμα να το φέρετε μαζί σας. Είναι ένα σημαντικό μήνυμα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ότι εστιάζουμε στα θετικά σημεία καταπολεμώντας τα αρνητικά. Είμαστε όλοι πολιτικοί. Και κατανοώ ότι και στα δικά σας εθνικά κοινοβούλια, όπως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι πολιτικοί εστιάζουν σε ένα θέμα όταν θεωρούν ότι το θέμα αυτό είναι πολιτικά χρήσιμο, όχι για τους ίδιους μόνο, αλλά είναι ένα θέμα στο οποίο υπάρχει ελπίδα, κάτι με το οποίο μπορούν να αλλάξουν κάτι. Κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί με κάτι που είναι χαμένη υπόθεση. Κανείς δεν θέλει ε, να ασχολείται συνέχεια με κάτι το οποίο καταραίει. Τα ανθρώπινα δικαιώματα λοιπόν δεν καταραίουν. Παρά τις προκλήσεις που υπάρχουν, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας. Μπορούμε να ασκούμε κριτική, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα εκατομμύρια των πολιτών σε ολόκληρο τον κόσμο που προσβλέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να ε, ενθαρρυνθούν. Υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία θα έπρεπε να είναι καλύτερα, αλλά για τον κόσμο, για ολόκληρο τον κόσμο, εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε αυτοί που κατάφεραν να βγουν από το αίμα και τον πόλεμο και το μίσος και να δημιουργήσουν ένα χώρο ευημερίας, της μεγαλύτερης ευημερίας σε ολόκληρο τον κόσμο σήμερα. Για αυτούς εμείς αντιπροσωπεύουμε το μέλλον τους. Ας μην τους ε, εγκαταλείψουμε λοιπόν, ας συνεχίσουμε να είμαστε εστιασμένοι σε αυτά τα οποία κάνουμε με αξιοπιστία, με ισχυρέ πεπιθήσει, κατανοώντα ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι χαμένη υπόθεση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην κοινωνία μας και στον κόσμο σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Κλείνουμε εδώ το πρώτο πάνελ και θα αρχίσουμε το δεύτερο. Τόκες μπορείς να με αντικαταστήσεις. Κυρίε Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φιλοξενούμενοι, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων, ας συνεχίσουμε. Έχουμε μείνει λίγο πίσω, έχουμε καθυστερήσει, πρέπει να είναι πιο σύντομες οι παρεμβάσεις. Εν είδη εισαγωγή να σας πω τα εξής. Moving now from the general κινούμεθα από το γενικό επίπεδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προς πιο συγκεκριμένο ειδικό τομέα. Θα εστιαστούμε επί των επιχειρήσεων και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ένα θέμα που συζητείται σε πολλά επίπεδα και σε πολλά βήματα συζητήσεων. Πολλοί φορείς εμπλέκονται στην προσπάθεια εξασφαλίσεως ότι ο επιχειρηματικός τομέας θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στα πλαίσια του διεθνούς τη διεθνού νομοθεσία στα ανθρώπινα δικαιώματα υπέχουν καθήκον τα κράτη-μέλη να διορθώσουν την κατάχρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιχειρήσει και όταν αυτέ κινούνται ακόμα και διασυνοριακά. Διάφορα εθνικά κοινοβούλια αντιμετωπίζουν κάποιες από τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συναφή ζητήματα μέσω θεσπίσεως νέας νομοθεσίας. Να αναφέρω κάποια κράτη. Εθνική Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας, το Ολλανδικό Κοινοβούλιο, ή η Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω υπάρχουν ε, διάφοροι κανονισμοί για ε, μη οδηγία για, μη, για, την, ε, για τα ορυκτά από περιοχή συγκρούσεων που πρέπει να υπάρχουν κάποιες συνθήκες που πληρούνται εταιρείε υλοτομίας, ξυλίας, που πρέπει να σέβονται σε τι εταιρείε τα εργατικά δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι παραβιάσει όμω ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τομέα τον επιχειρηματικών για να αντιμετωπιστούν χρειάζεται προσπάθεια από πολλά κράτη, όχι μόνο από ένα. Σε συγκεκριμένου τομεί, η διεθνή νομοθεσία απαιτείται για να εξασφαλίσει ότι οι εταιρείε θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όπου λειτουργούν. Να αναφέρω δύο πρωτοβουλίες του ΟΗΕ σχετικά με αυτό. Πρώτα, εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές για επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ, κάτι που υφετήθηκε το 2011. Εκεί αναφέρεται σαφώς ότι ο ιδιωτικός τομέας υπέχει ευθύνη να σέβεται και να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και να παρέχει αποζημιώσεις για τις και διορθωτικά μέτρα για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεξάρτητα από το αν είναι πρόθυμες οι κυβερνήσεις σε θέση να προστατεύσουν αυτά τα δικαιώματα. Δεύτερον, διακυβερνητική ομάδα εργασίας, διαρκής ομάδα εργασίας για την επεξεργασία ενός εργαλείου νομικά δεσμευτικού διεθνούς για ε, τις διεθνείς διασυνοριακές επιχειρήσεις ε, που πρέπει να σέβονται ανθρώπινα δικαιώματα. Και στόχος να υιοθετηθεί μια συνθήκη δεσμευτική κάποτε. Αυτή η ομάδα εργασίας συνεδρίαση για τέταρτη φορά από 15 με 19 Οκτωβρίου ε, τρέχοντος έτους. Στηρίζει την πολυμερή διαδικασία για να υπάρξει τελικά ένα νομικά δεσμευτικό εργαλείο όσον αφορά τις ε, ε, διεθνείς, τις τις ε, πολυεθνικές αυτές επιχειρήσεις και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτησε ένα ψήφισμα 4 ε, Οκτωβρίου φέτος για το πώς συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση του μέσου ε, του ΟΗΕ για αυτές τις επιχειρήσεις που θα πρέπει να σέβονται τα, τις υπερεθνικές που πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη είναι σε μοναδική θέση μπορούν να ηγηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την νομοθεσία και την πολιτική αυτή, ε, υιοθετώντα ε, όρους ε, στις επιχειρήσεις όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με την νομοθεσία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο πάνελ τώρα θα συζητήσουμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον επιχειρηματικό τομέα με ομιλητές από εθνικά κοινοβούλια εκπροσώπους συνδικάτων, εκπροσώπους του επιχειρηματικού τομέα, καθώς και ε, με τον πρόεδρο της ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για τη συνθήκη που επεξεργάζεται αυτή η ομάδα εργασίας, για αυτή τη συνθήκη που θα πρέπει να ετοιμαστεί, που θα είναι νομικά δεσμευτική. Καλωσορίζω την κυρία Μαχπουλέ Σαχά, διευθύντρια του νομικού τμήματο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων το γραφείο της επεξεργάζεται θέματα νομικά και θέματα πολιτικής που άπτονται των διεθνών προτύπων συνθήκων εργασίας. Έχετε το λόγο. Thank you very uh, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την εισήγηση και γιατί καλέσατε το ITUC, την ε, Διεθνή Συνομοσπονδία Συνδικάτων, να μιλήσει. Εκπροσωπούμε 207 εκατομμύρια εργαζομένων παγκοσμίω. Ε, μιλάμε για αξιοπρεπή εργασία και μία ε, σαφή αλυσίδα εφοδιασμού που είναι ύψης της σημασίας. Το τρέχον πρότυπο παγκοσμιοποίησης δυστυχώς λειτουργεί αντιθετικά. Οι, παγκόσμιες ε, ε, αλυσίδες, εφοδιασμού έχουν σαν ε, λόγο ύπαρξης την παροχή εφοδιασμού για όλους. Δυστυχώς όμως εδώ μιλάμε για ένα 10% των ε, επιχειρήσεων. Δυστυχώς, ένα 60% των, ε, του εργατικού δυναμικού μόνο έχει μια ουσιαστική σύμβαση. Οι μεγαλύτερες ε, 50 επιχειρήσεις δυστυχώς ε, ε, απασχολούν ένα 6% των εργοζομένων κατά αυτόν τον τρόπο. Τουλάχιστον ένα 94% του εργατικού δυναμικού βρίσκεται στην ε, παραοικονομία και γι' αυτό ε, δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με επισφαλή εργασία, με μισθούς ε, πείνας. Επίσης, δυστυχώς βρίσκουμε διάφορες μορφές ε, δουλεμπορίου, τα οποία ανέχονται στην εργασία. Φέτος και του χρόνου ιδιαίτερα η ΔΟΕ θα πανηγυρίσει το εκατοστό έτος ύπαρξης και γι' αυτό αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τις ε, δηλώσεις του Διεθνούς Γραφείου ή του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής δικαιοσύνης. Το 88% όμως των εργαζομένων δήλωσε στην ITUC ότι δυστυχώς δεν έχουν έναν επαρκή και διαφανή μισθό. Την προηγούμενη εβδομάδα ε, βρέθηκα στην έδρα της Αβίβα και είδα ότι δυστυχώς ούτε εκεί υπάρχουν benchmarks ε, για ε, σωστή μισθοδοσία. Ένα άλλο σημείο είναι ότι μόνο στο 3% των επιχειρήσεων έχουν ε, ληφθεί ένδικα μέσα για περίπτωση καταχρήσεων. Πιστεύω λοιπόν ότι έχει μεγάλη σημασία η χρήση των ένδικων μέσων, ιδιαίτερα στα πλαίσια του εταιρικού δικαίου. Οι πολυεθνικές εταιρείες δυστυχώς έχουν ένα μη διαφανές δίκτυο προμηθευτών και έτσι δεν υπάρχει λογοδοσία γιατί όταν υπάρχουν παραβιάσεις κανένας δεν λογοδοτεί. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν αποζητούν δικαιοσύνη κατά των εγχωρίων επιχειρήσεων μέσα στα πλαίσια των παροχών. Επίσης ε, ε, δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη ούτε στην παγκοσμιοποίηση αλλά ούτε και στις αρχές της δημοκρατίας. Η πλειοψηφία των ανθρώπων θέλουν να υπάρχει εγγύηση ως προς τα εργασιακά δικαιώματα. Οι 9 στους 10 θέλουν πιο αυστηρούς νόμους ως προς τις μεγάλες κοινοπραξίες που θα πρέπει να λογοδοτούν. Ως συνδικάτα θέλουμε να υπάρχει ελάχιστος μισθός και συλλογικές συμβάσεις καθώς και συλλογικές ε, διαπραγματεύσεις μέσα στα πλαίσια της παγκόσμιας κοινωνικής προστασίας. Όμως χρειαζόμαστε δράση και από την κυβέρνηση. Πολλοί εκπρόσωποι στο προηγούμενο πάνελ μίλησαν για, τον, ε, ε, για την υπέρ, υπέρ το δέον θεσμοθέτηση των ε, εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά θεωρώ ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο. Και χαίρομαι, διότι και άλλοι πάνελιστ ε, θα λάβουν το λόγο και χαίρομαι γιατί βρίσκεται μαζί μας και εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Εκουαδόρ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μέσα στα πλαίσια της ε, ε, δεοντολογίας έχουμε τον επόμενο ομιλητή που ασχολείται με τις ε, startups. Κύριε Κανό, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για την πρόσκληση και για να κάνω μία εισήγηση θα ήθελα να πω ότι εκπροσωπώ μια συμβουλευτική επιχείρηση που προσπαθεί να συνεργαστεί με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μέσα στα πλαίσια της τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα λοιπόν οι επιχειρήσεις να τηρούν αυτά τα δικαιώματα. Ε, έχω έχουμε εκπροσώπου σε πολλούς ε, τομείς, δηλαδή στον τομέα των επιχειρήσεων, του περιβάλλοντος, της ενέργειας και ούτω καθεξής. Προσπαθούμε λοιπόν να φτάσουμε σε έναν κώδικα δεοντολογίας έτσι ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να τηρούν το ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα λαμβάνουμε υπόψη μία πρακτική θεώρηση ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που εργάζονται στη Λατινική Αμερική. Θα ήθελα να πω ότι αυτή η παρουσίαση δεν αφορά τη γνωμοδότηση των επιχειρήσεων πελατών, αλλά τη δυνατότητα ταυτοποίησης των δυσκολιών και δυσχεριών, καθώς και των προκλήσεων που έχουμε και τη δράση των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων καθώς και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις αυτές. Θα ήθελα να πω ότι στην εφαρμογή αυτή ε, έχουμε μία αρχή που δεν έχει σχέση με τον υποχρεωτικό χαρακτήρα εφαρμογής των μέτρων. Έχουμε να κάνουμε με τέσσερις σε πέντε λόγους που σχετίζονται με την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πρώτη έχει, τη σημασία, ε, έχει σχέση με τη σημασία της αγοράς, την ε, κεφάλαια αγορά και το πώς αντιδρούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, σε αυτή την επιλεξιμότητα δράσης η κοινωνία της εργασίας αλλάζει διαδραστικά μέσα στα πλαίσια της ε, δράσης και των millennials. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτή η διαδραστικότητα και ο κανονισμός προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Αυτή είναι μία κινητήριος δύναμη και φυσικά ο συντονισμένος, η συντονισμένη δράση των ΜΚΟ που βοηθούν τις επιχειρήσεις επαγγελματικά για να κατανοήσουμε πώς γίνονται καταχρήσεις και μη τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι πρέπει να δράσουν ως προς την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολλές φορές ε, υπάρχει μία στρεβλή κατανόηση του θέματος. Υπάρχει ακτιβισμός ε, μέσα στις επιχειρήσεις που λειτουργεί ως μικιό εντός της επιχείρησης έτσι ώστε οι διαπραγματεύσεις να είναι σωστές. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι επιχειρήσεις είναι ένας δραστικός φορέας για να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές προκλήσεις και αυτό για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυσικά υπάρχει και η πολιτισμική διάσταση των επιχειρήσεων ως προς τους, ε, ε, τις οικονομικές προκλήσεις θα πρέπει πρώτον να έχουμε καλύτερες ε, πληροφορίες και αυτό σημαίνει ποιοτικές ε, πληροφορίες σε σχέση με τις επιχειρηματικές σειράξεις θα πρέπει να κατανοήσουμε όχι μόνο τις ε, καταχρήσεις, αλλά και τα διδάγματα που αντλούμε από αυτές. Στη Βραζιλία υπάρχει δυστυχώς μεγάλη ε, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, βλέπουμε ότι υπάρχει μία βελτίωση και στον τομέα της ε, υδροηλεκτρικής ενέργειας, αυτών των επιχειρήσεων δηλαδή στη Βραζιλία. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη διακυβέρνηση εκεί όπου λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι στο Μεξικό, στη Βραζιλία, στην Κολομβία, στην Αργεντινή θα πρέπει να δράσουμε άμεσα μέσα στα πλαίσια της ευαλωτότητας των επιχειρήσεων που θα πρέπει να κατανοήσουν καλύτερα τα διλήμματα που υπάρχουν. Και τέλος, θα πρέπει αυτές οι πληροφορίες ε, να είναι προσβάσιμες στις αγορές, δηλαδή να ξέρουμε ότι υπάρχουν καταχρήσεις και να ε, γνωστοποιηθούν ε, στις κεφαλαίες αγορές. Διαφορετικά δεν θα υπάρχει παρά συνέχεια των επενδύσεων, η οποία θα έπρεπε να σταματήσει όταν υπάρχουν καταχρήσεις και μη τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα υπερβολικά ε, κανονιστικό πλαίσιο. Ε, ένα λεπτό έχω ακόμα στη διάθεσή μου ίσως και να το έχω υπερβεί, αλλά θα ήθελα να πω ότι στις επιχειρήσεις υπάρχει και μία πολιτισμική διάσταση την οποία θα πρέπει να αλλάξουμε, δηλαδή να δούμε τι γίνεται με την συμμόρφωση. Ε, θα πρέπει να υπάρχει τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβασμός, ε, δηλαδή, πολλές φορές οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αποκρύψουν τις καταχρήσεις και δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιστραφεί. Αυτά θα είχα να πω εν συντομία. Σας ευχαριστώ κύριε Κάνου. Ο κύριος Ντομινίκ Πουατιέ, μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της ε, Γαλλική Εθνοσύνη Λέψο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Καλημέρα σε όλους. Είμαι πολύ ευτυχής που μπορώ να μιλήσω σήμερα την ημέρα που γιορτάζουμε τη διακήρυξη ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να σας πω τι έγινε στο τελευταία χρόνια στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση που οδήγησε στην περασμένη άνοιξη να θετηθεί ένας νόμος που σήμερα είναι πρωτοπόρα νομοθεσία ε, για, για τις ε, ε, για τις υπεργολαβίες, για τις παραγγελίες, τον έλεγχο αυτών κλπ. Έγινε μεγάλη μάχη που έγινε από έναν κύκλο, ηγηθήκανε ΜΚΟ, οι περισσότερες από αυτές, τα περισσότερα συνδικάτα τα γαλλικά, τα πανεπιστήμια συμμετείχαν και οι βουλευτές όσον αφορά τον πολιτικό τομέα ε, και οι περισσότεροι ανήκαν στην προηγούμενη θητεία, αλλά κάθε φορά συμμετείχαν βουλευτές ε, που ξέφευγαν από τα κόμματά τους στην προσπάθεια που κατέβαλαν. Ε, έγινε η μάχη παρά τις δισταγμούς του επιχειρηματικού κόσμου, παρά το συντηρητικισμό και τη νεοφιλελεύθερη τοποθέτηση, αλλά χάρη στις προσπάθειες του Κοινοβουλίου και της κοινωνίας των πολιτών τελικά θεσπίθηκε ε, η νομοθεσία και ήταν πραγματικά μια δημοκρατική νίκη για τη χώρα μας αλλά και για όλο τον κόσμο. Περί τίνος πρόκειται λοιπόν. Θέλουμε να, προ... να... όπως προτείνει ο ΙΕ και ο ΣΕ, ο ΣΑ μάλλον και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα να ειδοποιούμε όταν υπάρχουν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της νομοθεσίας περιβάλλοντος. Και τώρα πια αυτό είναι καινούριο. Οι παραβιάσει ε, τη νομοθεσία κατά του περιβάλλοντο ε, εξισούται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή, προστατεύουμε την αξιοπρέπεια τη ανθρωπότητα υπό την έννοια τη προστασία του ατόμου και τη προστασία του περιβάλλοντο για την προστασία του κοινού οίκου. Είναι κοινή μάχη και θα πρέπει το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η νομοθεσία να τα καλύπτει σε ίση βάση, ε, στο ίδιο δημοκρατικό πλαίσιο. Λοιπόν, ε, για πρώτη φορά λοιπόν αυτός ο νόμος ε, με καταναγκαστικό τρόπο ε, οδηγεί στην παρέμβαση ενός δικαστού στην εθνική επικράτεια στις περιπτώσεις της παραβιάσεως γίνεται μια αποκάλυψη για πρώτη φορά καταγγελία προβλέπεται μια καταγγελία μάλλον καθορισμός μεταξύ του εντολέα και του εκτελεστή της εντολής των αποστολών που εκτελούνται σε διάφορα σημεία είτε πρόκειται για αγαθά στον αγροτροφημικό τομέα, είτε πρόκειται για προϊόντα κατασκευαστικού τομέα, ηλεκτρονικών προϊόντων ή δημοσίων έργων. Η ευθύνη του εντολέα ε, καθορίζεται πλέον και χάρη σε ένα σχέδιο επαγρύπνησης. Δηλαδή, βάσει αυτού εντοπίζονται διάφοροι κίνδυνοι που αναλαμβάνει στον κόσμο μια επιχείρηση, αναθέτοντα την παραγωγή τη μέχρι και στην άλλη άκρη του πλανήτη. Υπάρχει χαρτογράφηση των κινδύνων και χρειάζονται τα δέοντα μέτρα, ώστε να αποφευθεί η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προστασία του περιβάλλοντο. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του περιβάλλοντο ε, με ρεαλιστικό τρόπο καλύπτονται με βάση τις αρχές του Τζον Ρούμπινγκ ε, για του ΟΗΕ αρχή που έχει θεσπιστεί σε όλα τα διεθνή βήματα Λοιπόν, αυτές οι αρχές διακυβεύονται. Θέλει η γαλλική νομοθεσία να εφαρμόσει σταδιακά, προοδευτικά αυτές τις αρχές πάνω στις μεγάλες επιχειρήσεις, 100, ε, δηλαδή 250 επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 100.000 μισθωτούς καλύπτονται σε πρώτη φάση, περίπου τα 2 τρίτα του εξωτερικού εμπορίου αντιπροσωπεύουν της χώρας μας είναι οι πιο ισχυροί που να δώσουν το παράδειγμα που ξεκινήσουν. Δεν είναι ασήμαντο ε, αυτό το ποσοστό. Οι πιο μεγάλε υπερεθνικέ, είτε είναι γαλλική προελεύσεω, ε, γαλλική καταγωγή ή που έχουν μια σημαντική δραστηριότητα των θηγατρικών του εταιριών στη χώρα μα, καλύπτονται. Λοιπόν, εγκαθιστά αυτή η νομοθεσία κατά κάποιο τρόπο ένα τρίτο δρόμο μεταξύ των ε, νομοθετικών συστημάτων που δεν είναι τόσο ρεαλιστικά όσον αφορά την πραγματικότητα των περιπλόκων αλυσίδων ε, διατροφής και απ' την άλλη ε, το, την ήπια νομοθεσία. Αυτά είναι τα δύο άκρα. Έχουμε τώρα μια τρίτη οδό, διότι η νομοθεσία που εφαρμόζεται από τις ε, εταιρείε βάσει της εμπειρογνωμοσύνης τους ε, και αυτή είναι η ισχύ της νομοθεσίας που κινητοποιεί τις επιχειρήσεις να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να ειδοποιούν για τους ε, κινδύνους που αντιμετωπίζουν και πρέπει οι εταιρείε να βρουν λύσεις. Ο, ο δικαστής πρέπει να κρίνει την αποτελεσματικότητα των λύσεων που εφαρμόζουν οι εταιρείε. Είναι μια καινοτομία νομοθετική που κινητοποιεί ε, τις εταιρείε και τελικά ε, οποιοδήποτε μπορεί να καταγγείλει μια επιχείρηση πολυεθνική η οποία δεν έχει εφαρμόσει το, σχέδιο επαγρύπνησης. Η τοπική αυτοδιοίκηση οποιοδήποτε φορέας αρμόδιος εδώ στην άλλο άκρο του κόσμου, θύμα, η ε, ΜΚΟ, συνδικάτα, κράτη, όλοι μπορούν να προσφύγουν σε Γάλλο δικαστή που θα αποφασίσει αν θα πρέπει να επιληφθεί. Μια επιχείρηση μπορεί να καταδικαστεί διότι δεν έχει ένα σχέδιο επαγρύπνησης ή κακό σχέδιο επαγρύπνησης και σε περίπτωση προβλημάτων σοβαρών, αν δεν έχουν κινητοποιηθεί τα μέτρα πρόληψης, το, σχέδιο, το, το να μην έχει ένα σχέδιο επαγρύπνησης είναι κάτι επιβαρυντικό για την απόφαση περί ποινών και αποζημιώσεων. Είναι πολύ καινοτόμα αυτή η προσέγγιση. Ξεπερνούμε το παραδοσιακό εμπόδιο της εξοδαφικότητας εγκαθιδρύοντας αυτό το μέτρο. Από μια μοναχική ε, ε, κυριαρχία πάμε σε αλληλέγγυα ε, τέτοια δικαιοδοσία. Το 2017 υιοθετήθηκε η νομοθεσία. Έχουν μπει σε περίοδο του επί μαθητείας 250 επιχειρήσεις στη Γαλλία μέχρι το τέλο του έτους και από 1η Πρώτου 2019 μια νομολογία μπορεί να καθεδρυθεί διότι ο νόμος αυτός θα ισχύει πλέον ε, και εμπνέει την ομάδα εργασίας του ΟΗΕ. Αυτή η νομοθεσία εμπνέει διάφορα κράτη Έχω πάει σε διάφορες πρωτεύουσε και κοινοβούλια και της Ευρώπης και τα συνδικάτα και διάφορα ερευνητικά κέντρα ενδιαφέρονται πολύ από την νομοθεσία. Και θέλω να κλείσω ότι ίσω ανήκει στις τρει-τέσσερι συναπόφαση των συγκαθορισμού της μυθολογίας, παραβίαση, ε, αποφυγή της φοροδιαφυγής. Μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή μπορούμε να δημιουργήσουμε τελικά ένα ευρωπαϊκό μοντέλο των επιχειρήσεων που να αποτελέσει μια πραγματική ε, δύναμη στην παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστώ κύριε Μπουατιέ, λέει ο πρόεδρο. Και τώρα ο κύριος Μανουέλ Αλτάβα, μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Πρόεδρος Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας από την Ισπανία έχει το λόγο. Muchas gracias. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Πώς ξέρετε τον Ιούνιο το 2014 ο Ισημερινός και η Νότιος Αφρική αποφάσισαν να λάβουν μια πρωτοβουλία για την κατάρτιση μιας ε, διεθνούς συμφωνίας ως προς την προστασία των επιχειρήσεων και των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην Ισπανία στις 28 Ιουλίου 2017 ε, ενεκρίθη το σχέδιο εθνικής δράσης επιχειρήσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στα πλαίσια των κατευθυντηρίων γραμμών των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι συμμετείχε η δημόσια διοίκηση, οι επιχειρήσεις και η κοινωνία των πολιτών κατά τη διάρκεια δύο ετών μετά από μία συνεχή εργασία που ε, συνεχίστηκε και τους τελευταίους μήνες. Θέλουμε λοιπόν να θέσουμε σε εφαρμογή τις αρχές που διέπουν τα Ηνωμένα Έθνη στις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με βάση το ψήφισμα που ενεκρίθη τον Ιούνιο του 2014, ψήφισμα 17,4 Άρα η Ισπανία θέλει να, να προσπαθήσει να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα τη στιγμή που επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττει ε, ακριβώς αυτά μέσα στα πλαίσια όλων των χωρών με τις οποίες συνεργάζεται. Θέλει επίσης να υπάρχει σχετικό προτέρημα των ε, ισπανικών επιχειρήσεων έτσι ώστε να μπορέσουν να δράσουν τηρώντας απόλυτα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το σχέδιο αποτελεί την απαρχή μιας διαρκούς διαδικασίας. Η διάρκεια του είναι τριετής μέχρι τον Ιούλιο του 2020 και έχει την κατάλληλη εργαλειοθήκη έτσι ώστε να παρακολουθήσει αυτή τη διαδικασία το Υπουργείο Εξωτερικών και η Ευρωπαϊκή Ένωση με συνεργασία της Ισπανίας θα θέσουν σε εφαρμογή αυτό το σχέδιο. Η Ισπανία λοιπόν προτίθεται να προωθήσει δράσεις ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα με υποστήριξη μέσω επιχορηγήσεων. Επίσης να προωθήσει τις επιχειρήσεις για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στα πλαίσια της ε, αναπτυξιακής συνεργασίας. Η εξωτερική μας, η υπηρεσία μας εξωτερικής δράσης ε, έχει ως ε, κύριο μέλημα την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις επιχειρήσεις. Αυτό αφορά και τις διπλωματικές υπηρεσίες, τη μόνιμη αντιπροσωπεία, τις μόνιμες αντιπροσωπείες και τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών καθώς και των κέντρων κατάρτισης. Και φυσικά αυτά μέσα στα πλαίσια της, ε, του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό αφορά και τις μεγάλες αλλά και τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις δρώντας κατά αυτόν τον τρόπο, το σχέδιο της Ισπανίας μετριάζει τις αρνητικές συνέπειες που απορρέουν από την ε, παγκοσμιοποίηση, ε, δημιουργώντας ανισότητες μεταξύ κρατών, κοινοτήτων, προσώπων και επιχειρήσεων όσον αφορά την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα στις πιο φτωχές γωνιές του κόσμου. Επίσης υπάρχει μία διακυβερνητική ομάδα των Ηνωμένων Εθνών για να οριστεί ένας, ε, μια δεσμευτική συμφωνία για να αντιμετωπίσει την ατιμορρησία των μεγάλων επιχειρήσεων. Επίσης ε, συμμετέχει και η κοινωνία των πολιτών κοινότητες, ε, φυσικά πρόσωπα και η ακαδημαϊκή κοινότητα με βάση τους ε, νόμους και τις αρχές που διέπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για να ορίσουμε μία μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να τηρηθούν ε, οι διεθνείς προδιαγραφές για τις διεθνείς επιχειρήσεις. Θα πρέπει να κινηθούμε πέρα από το εθελοντικό χαρακτήρα συνεργασίας. Θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός για να φτάσουμε σε ένα οικονομικό σύστημα που θα τηρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσώπων και την ευημερία τους και για να σταματήσουμε με την ε, ατιμορρησία των μεγάλων πολυεθνικών. Τέλος, πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ισπανία θα πρέπει να ορίσουν αυτό το μέσο το οποίο να είναι δεσμευτικό προς όλες τις επιχειρήσεις εθνικές ή πολυεθνικές έτσι ώστε τα κράτη και οι επιχειρήσεις να τηρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στα πλαίσια της δήλωσης των Ηνωμένων Εθνών. Σας ευχαριστώ. E ναι, και τώρα δίνουμε το λόγο ε, στην επόμενη ομιλήτρια, ε, εντεταλμένη της ε, αποστολής του Εκουαδόρ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να χαιρετήσω τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια, καθώς και τους πάνελιστ. Εξ ονόματος του Εκουαδόρ, σας ευχαριστώ που μας επιτρέπετε να σας μιλήσουμε για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις ως προς το Διεθνές Μέσο για την προστασία των εργαζομένων στις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Εμείς συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γνωρίζουμε ότι πολλά κράτη την έχουν προσυπογράψει. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας ε, ε, βασικός παράγων μέσα στα πλαίσια της δράσης των πολυεθνικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν βέβαια, υπάρχει και μη δεσμευτικό πλαίσιο, όμως ε, η πείρα καταδεικνύει ότι δεν μπορούμε να παραμείνουμε σε αυτό το πλαίσιο. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτό το δεσμευτικό μέσο είναι αναγκαίο για να υπάρχει σωστή μεταχείριση των ε, θυμάτων παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρακαλώ να μιλάτε λίγο πιο αργά, προτρέπει ο Πρόεδρος. Ε, επιπλέον ένα 80% των αγαθών και υπηρεσιών παράγονται μέσα από μια κατακαιρματισμένη παραγωγή η οποία δεν ε, ε, τηρεί τα σύνορα και δεν λαμβάνει υπόψη δηλαδή τα εθνικά σύνορα. Γι' αυτό τον Ιούνιο του 2014 το Εκουαδόρ και η Νότια Αφρική προετοίμασαν το ψήφισμα 26,9 της 26ης ε, διάσκεψης του Συμβουλίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, έτσι ώστε να προωθηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ως προς τη δράση των πολιεθνικών. Σύμφωνα με την πρακτική του Συμβουλίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Εκουαδόρ θα πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία. Από το 2015 έχουν γίνει τέσσερις συνεδριάσεις, η τελευταία τον προηγούμενο Οκτώβριο, γιατί για πρώτη φορά λειτουργήσαμε με βάση ένα προσχέδιο με 15 άρθρα. Η πρώτη ανάγνωση του δεσμευτικού μέσου έγινε ε, υπό, τη, υπό τον ύπατο εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών. Το κείμενο ε, συμπεριλαμβάνει βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως τις βασικές ε, ευθύνες και καθήκοντα κρατών και επιχειρήσεων. Το προσχέδιο αυτό δεν δημιουργεί νέες υποχρεώσεις, αλλά εγγυάται την εφαρμογή αυτών που προϋπάρχουν μέσα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, ιδιαίτερα εκεί που υπάρχουν νομικά προσκόμματα, ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να μην αντιδρούν και να μην αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους. Αυτή είναι μία βάση διαπραγμάτευσης η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί. Προβλέπονται τέσσερις βασικοί άξονες. Πρόληψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου, το δικαίωμα των θυμάτων να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η διεθνής συνεργασία για την πραγματική εφαρμογή του μέσου, καθώς και διεθνείς μηχανισμοί ελέγχου. Η σημασία της πρώτης ανάγνωσης του προσχεδίου έγινε υπό την παρουσία 95 εκπροσώπων κρατών ε, των ε, Ηνωμένων Εθνών και με τη συμμετοχή 400 εκπροσώπων της ε, κοινωνίας των πολιτών και ακαδημαϊκών. Επίσης, διεθνείς και εθνικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συμμετείχαν επίσης, συμμετείχε και η Εκκλησία με εκπροσώπους της, καθώς και ΜΚΟ που συνεργάζονται με το ε, Διεθνές Συμβούλιο Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών. Ε, θα πρέπει να μιλήσουμε για τη συμμετοχή 30 εμπειρογνωμόνων από όλες τις περιοχές του κόσμου που σχολίασαν τα άρθρα του προσχεδίου μεταξύ των συστάσεων και των συμπερασμάτων, καλούμε όλα τα κράτη-μέλη να υποβάλουν τα σχόλια και προτάσεις τους στο προσχέδιο αυτό μέχρι τα τέλη του Φεβρουαρίου του 2019 ως προς τη βάση των συζητήσεων κατά την τέταρτη σύνοδο της ομάδας εργασίας θα αναμένουμε τα σχόλια όλων μέχρι τον επόμενο Φεβρουάριο. Και ο πρόεδρος εισηγητής θα παρουσιάσει μία αναθεωρημένη έκδοση του δεσμευτικού μέσου που θα πρέπει κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει μέχρι τον Ιούνιο του 19. Η πέμπτη σύνοδος της ομάδας εργασίας θα ασχοληθεί με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβερνήσεων καθώς και το ε, βασικό πρωτόκολλο εθελούσια συνεργασίας. Στην, ε, μάλλον πριν από την Πέμπτη Σύνοδο θα γίνουν άτυπες ε, συναντήσεις με τα κράτη των Ηνωμένων Εθνών, ε, διακυβερνητικών οργανώσεων, μηχανισμών των Ηνωμένων Εθνών και επίσης άτυπες συναντήσεις μέσα στα πλαίσια του προγράμματος εργασίας εν ώψη της Πέμπτης Συνόδου. Γνωρίζουμε ότι αυτή η διαδικασία θα χρειαστεί πολλά χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί. Χρειάζεται ευρεία συνένεση και συμμετοχή για συγκεκριμένες δράσεις, συνενετικές δράσεις. Εάν η κοινωνίες συνδέονται περισσότερο μεταξύ τους, τότε θα μπορέσουμε να ορθώσουμε το ανάστημά μας ως προς την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. And, ε, Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα μπορούν να έχουν το λόγο οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων. Έχουμε ήδη τέσσερις εγγεγραμμένους με χρόνο ομιλίας. Θα ξεκινήσω λοιπόν με αυτούς τους τέσσερις πρώτους. Καταρχήν, ο κύριος Βακελάρντε Βασκονσέλος από την Πορτογαλία. It is not ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα την ε, δυνατότητα τον Οκτώβριο να συμμετάσχω σε μία πρωτοβουλία της Αυστρίας στη Βιέννη που είχε ως θεματική την ε, παγκόσμια διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πώς εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη. Μιλήσαμε λοιπόν για τις δυσχέρειες που υπάρχουν για την σωστή νομική εφαρμογή των ε, προδιαγραφών της διακήρυξης αυτής. Και φυσικά το βασικό μας μέλημα είναι η καθημερινή ζωή και η εφαρμογή της διακήρυξης παντού. Αυτό που έχει σημασία είναι η διασφάλιση της καθολικότητας της διακήρυξης και η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αδιέρετη δηλαδή εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. δηλαδή να μην μιλάμε μόνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά ε, καθήκοντα και δικαιώματα, αλλά να δούμε πώς οι εθνικές δικαιοδοσίες μπορούν να εφαρμόσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή στις υποθέσεις που απασχολούν τα δικαστήρια. Βλέπουμε ότι δυστυχώς παρά το δεσμευτικό χαρακτήρα πολλές φορές ο δικαστικός τομέας δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Άρα και ο ίδιος ο προϋπολογισμός και το δημοσιονομικό πλαίσιο θα έπρεπε να λάβει υπόψη έμπρακτα την εφαρμογή της παγκόσμιας διακήρυξης. Ο πληθυσμός έχει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκαταλήψεις που έχει δημιουργήσει η παγκοσμιοποίηση. Μέσα στα πλαίσια του άκρα του καπιταλισμού και δυστυχώς μέσω των πολιτικών λιτότητας ε, κατεστάλησαν αυτά τα δικαιώματα όπως βλέπουμε και με τη λυπηρή και πονίδι στη πολιτική που εφαρμόστηκε κατά της Ελλάδας. Άρα θα πρέπει να δούμε αυτή την αδιέρετη αρχή εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός. Ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος ομιλητής Μανώλη Πέτρο Φλωρίν. Σα ευχαριστώ πολύ. Έγινε λόγο για τι ανισότητες και τα ανθρώπινα δικαιώματα στον επιχειρηματικό κόσμο. μα. ενδιαφέρουν λοιπόν τα δικαιώματα πρωτίστως των εργαζομένων. Είναι σωστή αυτή η θεώρηση, αλλά ανεπαρκής, γιατί θα πρέπει να δούμε ποιοι αποκλείονται από την αγορά εργασίας γιατί δεν συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό σύστημα όπως θα έπρεπε. Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο ισχύει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός αυτής. Αφορά τους Ρωμά. Η απασχόλησή τους ε, είναι, ε, δεν, δεν έχει σωστή εφαρμογή. Και αυτό σας το λέω και ως ε, βουλευτής, αλλά γιατί είμαι και εγώ Ρωμά. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να καταβάλουν μία προσπάθεια να καταπολεμήσουν αυτές τις προκαταλήψεις και αυτό αφορά τις μεγάλες πολυεθνικές. Μερικές αντιμετωπίζουν το θέμα, αλλά η πλειονότητά τους όχι. Γι' αυτό νομίζω ότι η μεγάλη πρόκληση θα ήταν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συνεργαστούν ε, με τις πολυεθνικές για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα όσον αφορά τις ομάδες που αποκλείονται από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστούμε τον Πέτρε Φλωρίν. Ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Νόρντοβης, Ράσνους. από τη Δανία. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη για την ε, λάθος προφορά του ονόματός σας. Δεν πειράζει καθόλου, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ όλους ε, όσους έλαβαν το λόγο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις. Ε, παρακολουθώ τη δουλειά που γίνεται και στη Γαλλία, Αυτό που μας περιγράψατε, κύριε Ποτιέ και προσπαθούμε και στο Κοινοβούλιο στη Δανία να εφαρμόσουμε κάτι παρόμοιο. Είναι ένας αγώνας στον οποίο ε, προσπαθούμε να φέρουμε εις πέρας. Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε το παράδειγμα της Γαλλίας ή άλλων χωρών για να πούμε «Κοιτάξτε τι έχει γίνει σε άλλες χώρες». Και τώρα Είμαστε σε μια εποχή που χρειαζόμαστε περισσότερα νομικά δεσμευτικά εργαλεία και λιγότερα λόγια. Γιατί έχουμε κατευθυντήριε γραμμέ, αλλά όταν έχουμε επιχειρήσει ε, που μερικέ φορέ είναι μεγαλύτερε από κάποιε μικρέ χώρε, τότε το πρόβλημα μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. και η ομάδα εργασία ε, για νομικά δεσμευτικά εργαλεία για τι επιχειρήσει και τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, εκτελεί πολύ σημαντικό έργο. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μα τα εθνικά κοινοβούλια, τα ψηφίσματα αυτά τα γνωρίζω. Γνωρίζω το ψήφισμα που πέρασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά μετά τι γίνεται στην πράξη από το κράτο μέλο. Είναι πολύ πενιχρή η εφαρμογή σε επίπεδο κράτους μέλους. Στην κυβέρνηση στη Δανία προσπαθήσαμε να τους ε, πείσουμε να έρχονται στις συνεδριάσεις στην ομάδα εργασίας. Δεν ε, είχαμε καν αυτό διασφαλίσει. Τώρα θέλουμε να έχουμε νομικά δεσμευτικά εργαλεία, γιατί πέρασε ο καιρός για τα λόγια και για τις κατευθυντήριες γραμμές. Θέλουμε να περάσουμε στα έργα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και ο επόμενος ομιλητής, η επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Ελένη Σαμαγιάκη από την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κυρίες και κύριοι, ε, το Δεκέμβριο του 2000 υπογράφηκε στην Ίκαια της Γαλλίας ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων βάσει του οποίου τα εργασιακά δικαιώματα προστατεύονται ως ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα με βάση τις διατάξεις του χάρτη προστατεύεται το δικαίωμα στην εργασία, απαγορεύεται η αναγκαστική εργασία, προστατεύεται η συνδικαλιστική ελευθερία, το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση, απαγορεύεται η παιδική εργασία και προστατεύονται οι νέοι εργαζόμενοι και προστατεύεται η ισορροπία ανάμεσα στην οικογένεια και την επαγγελματική ζωή με ρητή αναφορά στη μητρότητα. Στην ελληνική νομοθεσία απαγορεύεται ρητά κάθε μορφή άμεσης ή έμεσης διάκρισης λόγω φύλου. Κάθε πρόσωπο προστατεύεται από την απόλυση για λόγους που συνδέονται με τη μητρότητα, καθώς και το δικαίωμά του να αμείβεται με άδεια μητρότητας ή γονική άδεια μετά τη γέννηση ή την υιοθεσία του παιδιού. Επιπλέον, άδεια για την ανατροφή του παιδιού μπορεί να πάρει ο πατέρας, ώστε να μην επομίζονται μόνο οι γυναίκες στην ευθύνη της μητρότητας. Πριν από μερικές μέρες, με νέες διατάξεις, το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης της Ελλάδας ε, καθιερώνει ειδικέ άδειε μητρότητας, τοκετού, λοχίας, εθυλασμού και φροντίδας του παιδιού. Δυστυχώς, οι διατάξεις αυτές δεν ισχύουν για τις ομογενοϊκές οικογένειες, δεν απολαμβάνουν δηλαδή τα ίδια δικαιώματα, αφού δεν έχουν αναγνωριστεί το δικαίωμα τεκνοθεσίας σε ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Με αποτέλεσμα ένας από τους δύο γονείς νομικά να είναι κατοχυρωμένος. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ε, αρκετές εθνικές και ενωσιακές ε, ε, συνθήκες και νόμοι που εξασφαλίζουν ε, τα δικαιώματα των εργαζομένων. παρόλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλές παραβιάσεις των δικαιωμάτων αυτών. Ε, ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφερθώ στο γεγονός ότι πολλοί εργαζόμενοι σε θέσεις χαμηλής ειδίκευσης εργάζονται σε έντονους ρυθμούς ενώ ταυτόχρονα αναφέρουν χαμηλά επίπεδα αυτονομίας και ανασφάλεια ως προς τη διατήρηση της θέσης τους και την ικανότητά τους να εργαστούν ξανά σε περίπτωση απόλυσης. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για εργαζόμενους ε, σε καθεστώς εργολαβίας. Σας είναι γνωστή η περίπτωση της Ευρωβουλευτή της κυρίας Κωνσταντίνας Κούνεβα η οποία δέχτηκε δολοφονική επίθεση όταν ήταν εργαζόμενη και μαχητική συνδικαλίστρια στο Σωματείο Καθαριστριών. Η κυβέρνηση της Ελλάδας με νόμο από το 2015 ε, και με μια σειρά από διατάξεις προβλέπει τη σύναψη ατομικών συμβάσεων έργου ε, ξεκίνησε μια διαδικασία να βάλει τέλος στο καθεστώς αυτό των εργολαβιών. Ε, μάλιστα δικαιώθηκε από πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που πρέπει να εφαρμοστούν όλα τα μέτρα για τα δικαιώματα ε, των εργαζομένων. Ε, στα πλαίσια αυτά, όταν μιλάμε λοιπόν για ανθρώπινα δικαιώματα και επιχειρήσεις, πρέπει να μιλάμε για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων, των γυναικών, των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, των ατόμων με αναπηρία, των νέων εργαζομένων, των εργαζομένων και των άνεργων άνω των 50 ετών, το δικαίωμα των μεταναστών και των προσφύγων στην εργασία, αλλά και για την προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων εντός και εκτός των εργασιακών χωρών. Ευχαριστώ πολύ. Last but not least, uh, Και τελευταίος τελευταία ομιλήτρια μάλλον, η κυρία Ρόζη Άλντα από την Ισπανία. Ε, Γεια σας και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμμετάσχω σε αυτή την υποεπιτροπή. Θα ήθελα να πω ότι στην τέταρτη ομάδα εργασίας, στη διακυβερνητική, στις 15 με 19 Οκτωβρίου ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχε επικοδομητικά σε όλες τις ομάδες εργασίας. Επίσης έγινε λόγος και για τα θύματα αυτής της ε, ευάλωτης εργασίας. Έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει συμμετοχή των θεσμικών εθνικών οργάνων έτσι ώστε να, ακουστούν οι φωνές, να ακουστεί η φωνή των θυμάτων μέσα στα πλαίσια της επιχειρηματικής δράσης. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο υπάρχουν ουσιαστικοί μηχανισμοί αποζημίωσης των θυμάτων. Ε, Ευχαριστούμε. Θα ήθελε κανείς άλλο το λόγο. Εσείς εκ μέρους των μη κυβερνητικών οργανώσεων, σωστά? Ήδη έχω δύο ονόματα. Η κυρία Αντριάννα Εσπινόζα, υπεύθυνη πολιτικής από τον Ευρωπαϊκό Συναστισμό Εταιρικής Δικαιοσύνης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα όλου του προλαλήσαντε και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι μία από τι βασικέ προκλήσει σήμερα είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε το σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην επιχειρησιακή λειτουργία των επιχειρήσεων παγκοσμίω. Και τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων συμβαδίζουν σε αυτή την προσπάθεια σήμερα. Θέλω να τονίσω ότι έχουμε εδώ μία μοναδική ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή. Ε, το, ο γαλλικός νόμος που ανέφερε ο κύριος Ποτιέ για το καθήκον επαγρύπνησης ε, ε, έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, αλλάζει την κατάσταση γιατί για πρώτη φορά υποχρεώνει τις μεγάλες εταιρείε να επιβλέπουν για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις δραστηριότητές τους και σε άλλες χώρες. Δεν είναι όμως μόνη χώρα η Γαλλία που εφαρμόζει κάτι τέτοιο σήμερα. Ήταν η πρώτη, αλλά σήμερα και άλλες χώρες αρχίζουν να εξετάζουν τέτοια νομοθετικά μέτρα που θα υποχρεώνουν τις εταιρείε ε, να ελέγχουν την αλυσίδα εφοδιασμού τους. Απαιτείται λοιπόν από εταιρείε ε, να εφαρμόζουν τη δέουσα επιμέλεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις ε, εταιρείε της, αλυσίδας, της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Ε, θα σας δώσω τρία παραδείγματα. Στην Ελβετία υπάρχει μια νομοθετική διαδικασία για υποχρεωτική νομοθεσία, για δέουσα επιμέλεια στα ανθρώπινα δικαιώματα και υπάρχει μεγάλη υποστήριξη και από την κοινωνία και από τις επιχειρήσεις. Η Ολλανδία και η Αυστρία επίσης εξετάζουν ε, τέτοια θέματα για την παιδική εργασία και η γερμανική κυβέρνηση έχει εξετάσει το ενδεχόμενο ε, νομοθετικών διατάξεων για την δέουσα επιμέλεια στα ανθρώπινα δικαιώματα από εταιρείε. Αυτό το οποίο κάνουν λοιπόν οι χώρες αυτές είναι ότι ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη φωνή της κοινωνίας που ακούγεται και ζητάει κάτι τέτοιο γιατί ε, όλο και περισσότερο η κοινωνία ζητάει να σέβονται οι εταιρείε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκστρατείε στο Λουξεμβούργο, στη Φινλανδία και αλλού ε, κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Η νομοθεσία αυτή λοιπόν για τη δέουση επιμέλεια στα ανθρώπινα δικαιώματα έχει υποστήριξη από όλε τι πλευρέ, διότι θα ε, αποφεύγει παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων και θα προσφέρει και ε, επανόρθωση για την περίπτωση παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολύ σημαντική λοιπόν αυτή είναι η νομοθεσία. Επομένως ήδη βρισκόμαστε στο σημείο της αλλαγής Η κοινωνία των πολιτών και οι εταιρείε ε, καθοδηγούν ε, την πορεία αυτή σε πολλά κράτη-μέλη και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το κίνημα προς μια περισσότερο βιώσιμη οικονομία αποδεχόμενη και υιοθετώντα τέτοια νομοθεσία για τα δικαιώματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εταιρείες. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντέμπι Στότχαρτ, συντονίστρια του δικτύου ΑΣΕΑΝ για τη Βερμανία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκπροσωπώ και την PDS. Επιτόπου εργάζομαι κοντά στον κόσμο στην Ασία. Και τι βλέπουμε ότι η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με επιχειρηματικέ δραστηριότητε γίνεται ένα από τα πιο σοβαρά φαινόμενα, από τι πιο σοβαρέ επιτόπιε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκτιμούμε πολύ το ότι εστιάζεσαι από αυτού. Ακόμα και στο Μιανμάρ, όπου έχουμε τη γενοκτονία των Ραχίνγκα, εκεί βρίσκουμε ότι υπάρχει οικονομική και επιχειρηματική διάσταση στην κρίση. Όσον αφορά τις κατεδρίες γραμμές για επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα το ΙΕ, είναι εξωσημείωτο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια δεν έχει ένα σχέδιο δράσης περιφερειακό για τις επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα και η παρούσα Προεδρία, η Αυστρία, ακόμα δεν έχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης, ούτε η Ρουμανία που θα αναλάβει την επόμενη Προεδρία του χρόνου. Αλλά νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να κάνουμε ένα άλμα και να ξεπεράσουμε τις εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές και να περάσουμε στη θέσπιση ενός μοντέλου, όπως ε, το νόμο για τη συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα που εφαρμόζει η Γαλλία και θα πρέπει να ακολουθήσουμε την ηγεσία του Εκουαδόρ όσον αφορά τη δουλειά που έχει γίνει εκεί σε διακυβερνητική ομάδα στον ΟΗΕ για νομικά δεσμευτική συνθήκη, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε το ότι οι επιχειρήσει θα πληρούν τι υποχρεώσει του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει να δώσουν δυνατότητα στι χώρε που θα προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα να μπορέσουν να τα προστατεύσουν στην επικράτειά τους. Θέλω να πω επίσης ότι δυστυχώς έχοντας πάει στη Γενέβη στα, στα περιθώρια της συνεδριάς της κυβερνητικής ομάδας για δεσμευτική ε, συμφωνία, είδαμε απογοήτευση ότι ήταν, ε, δημιουργούσε εμπόδια η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά αυτή τη νομικά δεσμευτική συνθήκη. Και αυτό δεν ταιριάζει καθόλου με τις αξίες της Ευρώπης και τις δηλωθήσεις αξίες ε, και την επιθυμία που έχει εκφράσει το Ευρωκοινοβούλιο. Εκτιμούμε το επιτελεστέν έργο διαφόρων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που επιδιώκουν πλήρη και συνεκτική εφαρμογή των υποχρεώσεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στα πλαίσια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Πρέπει να πω ότι όσον αφορά το εμπόριο και τις επενδύσεις και τις σχετικές συμφωνίες δεν είμαστε πλέον στις Βρυξέλλες, είμαστε στην Άγρια Δύση, είμαστε καουμπόιδες. Γιατί το λέω αυτό, διότι το 2016 ο Συνήγος του Πολίτη θεώρησε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένοχη για κακή διαχείριση. Ε, δεν μπόρεσε να κάνει πρώτερη αξιολόγηση αντικτύπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα Συμφωνής Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιετνάμ. Δύο χρόνια αργότερα, φέτος, η Συμφωνία για Προστασία Επενδύσεων Ευρωπαϊκής Ενώσεως Βιετνάμ συγκλονίζει διότι δεν παρέχει προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε ότι το τελευταίο 18 μήνο οι αρχές του Βιετνάμ ξεκίνησαν ε, μία από τη μεγαλύτερη καταπίεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων της τελευταίας δεκαετίας. Αν θέλουμε να δούμε να υπάρχει συνέπεια και συνοχή όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πολιτική, πρέπει να έχουμε μια γενική αναδιάθρωση της διαδικασίας και του περιεχόμενου των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου και των συμφωνιών προστασίας επενδύσεων. Θα κλείσω με πολύ μεγάλη επίκριση του ISDS ε, το μηχανισμό διευθετήσεως διαφορών για τους επενδυτές. Είδαμε ότι έχει αποτελέσει αντικείμενο κατάχρηση για να προστατεύσει τι εταιρείε και να επιτρέψει τι εταιρείε να αποφύγουν τι υποχρεώσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αποζημιώσει σε πληγήσει κοινότητε. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Όταν αρχίζουμε μια εταιρεία να λέει ότι πρέπει να έχει το δικαίωμα να μην πληρώνει για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να επενθυμίσουμε ότι όταν η δουλεία καταργήθηκε στην Ευρώπη, οι έμποροι δούλων αποζημιώθηκαν για απώλεια κερδών από το εμπόριο από το δουλεμπόριο. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μια επανάληψη αυτής της παράδοσης σε αυτή την περιοχή και στον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, άλλον έναν βουλευτή έχουμε που επιθυμεί να μιλήσει. Αλμπέρτο Αϊρόλα μέλος του Ιταλικού Κοινοβουλίου. Έχετε το λόγο. Ε, καλημέρα, ευχαριστώ. Είμαι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που μόλις ε, δημιουργήθηκε. Σημερίζομαι πλήρως αυτό που κάνει η Γαλλία όσον αφορά τις ευθύνες των, των ε, πολυεθνικών εταιριών που δεν σέβονται τη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτά που είπε ο Πορτογάλος συνάδελφος που κατά κάποιο τρόπο όπως είπε και ο Δανός συνάδελφος πρέπει να περάσουμε από προσανατολισμούς και σε χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μέσα πιο δεσμευτικά ευπρόσδεκτα τα δεσμευτικά μέσα Συχνά το πρόβλημα που διαβλέπω είναι το εξής, ότι σε σχέσεις μεταξύ πολυεθνικών και χωρών κυρίως της Αφρικανικής Υπήρου υπάρχουν σοβαρότατες περιπτώσεις παραβιάσεως των οικονομικών δικαιωμάτων και κατά συνέπεια ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως κάποια ορυχεία, εργάτες που εργάζονται σε πολύ κακές συνθήκες, όπου οι πολυεθνικές, οι χώρες που εμπορεύονται, που αποκτούν αυτά τα προϊόντα, ε, εθελοτυφλούν, στρέφουν αλλού το βλέμμα. Δε, δεν είναι μόνο σημαντικό να πλήττονται οι πολυεθνικές που διαπράττουν αδικήματα ή δεν σέβονται τους κανόνες. που δεν σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά χρειάζεται και έργο εντός των, του ΟΗΕ όπου εκεί δρεύουν οι ίδιοι πρόεδροι που επιτρέπουν στις χώρες τους να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα να δημιουργούνται καταστάσεις ε, δουλεία στην πράξη όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας. Πρέπει να υπάρξει μία προσπάθεια με συμμετοχή εκεί, αλλιώς πλήττουμε μόνο τις πολυεθνικές. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι δεν θα εργαστεί μία πολυεθνική σε κάποια συγκεκριμένα πλαίσια, αλλά όταν είμαστε στον ΟΗΕ έχουμε δίπλα μας ενδεχόμενα υπευθύνους για πολύ σοβαρές παραβιάσεις. Άρα είναι σημαντικότατο να ενεργοποιηθούμε και σε αυτό το μέτωπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να προσθέσω, αγαπητό ακροατήριο, αγαπητοί συνάδελφοι, και για τα νέα μέλη της Ένωσης, ούτως υπήν, χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό, σοβαρή πρόκληση. Η σχέση μεταξύ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επενδύσεων, οι πολυεθνικές εταιρείες που μετά την ολοκλήρωση, την ένταξη των χωρών, ήρθαν στις χώρες μας και υπάρχουν πολλές εντάσεις και αδικίες σε αυτό το τομέα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρόβλημα εντός της Ένωσης. Όχι μόνο σε τρίτες χώρες του κόσμου. Τέλος, να δώσω το λόγο για ένα, ενάμιση λεπτό σε σας που συμμετείχατε στο πάνελ με την ίδια σειρά. όπως όταν ξεκινήσαμε. Η κυρία, Σάχα, κυρία Σαχάν έχει το λόγο πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα σχόλιά σας ευπρόσδεκτο αυτό να σταματήσει ο παγκόσμιος καπιταλισμός, αυτό που μας είπε ο Πορτογάλος εκπρόσωπος. Τι ζητούμε, μια μεταμόρφωση του μοντέλου εφοδιασμού που να δουλέψει και για τους εργαζόμενους. Ευχαριστώ και την Ελληνίδα εκπρόσωπο που εύγλωτα περιέγραψε τι εννοούμε με τους εργαζομένους. Δεν είναι μόνο ε, ε, είναι εκείνοι που προσπαθούν να βρουν δουλειά, όχι μόνο αυτοί οι εργαζόμενοι που ε, εργάζονται με σε εργασία που χρειάζεται πολλέ γνώσει, αλλά και του ευάλωτε ομάδε, αυτού που εργάζονται με επισφαλεί συνθήκε κλπ. Άρα χρειάζεται να καλυφθεί ευρύ φάσμα εργαζόμενων. Πολύ ενθαρρυντικό που ακούσαμε ότι οι διάφοροι βουλευτέ εμπνέονται από την ομοθεσία τη γαλλική δείχνει ότι εξακολουθούν να έχουν κέρδη οι γαλλικέ εταιρείε. Ελπίζω να συνεχίζουν να τα μοιράζονται με του εργαζομένου που προξενούν τα κέρδη. Δεν κατέρευσε η γαλλική οικονομία. Είναι δίκαιο να πούμε ότι το να ζητάμε από τι εταιρείε να λάβουν προληπτικά μέτρα δεν πρέπει να θεωρηθεί κάτι τόσο ριζοσπαστικό σαν απέτηση. Όλοι θα πρέπει να ζητήσουμε να τεθεί τέρμα στο ανταγωνιστικό όφελος που έχουν κάποιες εταιρείε επειδή δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και εκείνες που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Άρα χρειαζόμαστε ε, ισότιμες συνθήκες εργασίας. Αυτές πρέπει να δημιουργηθούν. Απηχώ και εγώ αυτά που είπε η καλή μου φίλη Βίκη. Θέλουμε να ακούσουμε όλες τις φωνές και τις δικές σας φωνές και συζητήσεις για τη συνθήκη του ΟΗΕ ανταλλάσσονται απόψεις και έγινε μια πάρα πολύ καλή ανταλλαγή των πρακτικών και ελπίζω και την επόμενη φορά να ακούσουμε πολλά περισσότερα από σας. Ευχαριστώ. Κύριε Σανό. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα όλες τις παρεμβάσεις. Φυσικά χρειάζονται πιο δεσμευτικές συμφωνίες και αυτό αφορά ιδιαίτερα τον ιδιωτικό τομέα γιατί οι επιχειρήσεις είναι οι κόκκινες γραμμές της υλοποίησης. Μιλήσαμε και για την παγκόσμια διακυβέρνηση. Θα πρέπει να δούμε ποιες ε, ε, χώρες έχουν ε, το κατάλληλο προβάδισμα ως προς την τήρηση του δεσμευτικού χαρακτήρα. Μιλάμε για, ελάχιστες, για τις ελάχιστες ε, προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρηθούν ε, παντού ως προς την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλές ε, φορές θα πρέπει να δούμε και την περίπτωση της Γαλλίας, Γερμανίας και Ισπανίας, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και ευθύνη τα ανθρώπινα δικαιώματα στον επιχειρηματικό κόσμο θα πρέπει να αποτελέσουν ε, χρηστή πρακτική που να απορρέει από τα κοινοβούλια. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι οι επιχειρήσεις έχουν αλλάξει δρόμο και αυτό που έχει σημασία να δούμε και τις αρνητικές αλλά και τις ε, θετικές ε, απόρριες και συνέπειες και τη δράση των μίκιο, Να δούμε δηλαδή και την διαδικασία μεταφοράς αυτού του υποχρεωτικού πλαισίου. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Πουατιέ από την Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή. Πολύ ανέφεραν το ρυθμό που πρέπει να ακολουθήσουμε για να υιοθετήσουμε ε, τις ε, κατάλληλες αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύω ότι πρέπει να επιταχύνουμε γιατί οι συνθήκες είναι επικίνδυνες και ε, είναι παράγον ειρήνη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι και παράγον για την καλύτερη ανταγωνιστικότητα γιατί η ανταγωνιστικότητα στο μέλλον περνάει από την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι θα κερδίσει η Ευρώπη. Δεν θα κερδίσει με άλλους τρόπους αλλά θα νικήσει στην οικονομία του μέλλοντος εάν υιοθετήσει σαφώς τις αρχές που υιοθετήσαμε στη Γαλλία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όχι λοιπόν ημίμετρα, όχι δισταγμό, και για την εργασία των παιδιών και για όλα τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να υιοθετήσουμε αυτέ τι γενικέ αρχέ. Και τα καλά νέα ότι είναι ότι οι γενικέ επιχειρήσει έρχονται και με επισκέπτονται και μου λένε ότι με αυτό το σχέδιο υπαγρύπνηση έχουν μια νέα δυναμική, έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτή τη νέα δυναμική γιατί είναι η δυναμική του μέλλοντο. Την ίδια δυναμική είδαμε και για την καταπολέμηση τη δουλεία το 18ο αιώνα την ίδια αντίσταση είχαμε συναντήσει και για ε, την νομοθεσία για τα ατυχήματα στον εργασιακό χώρο. Κάθε φορά που υπήρχαν ε, ε, κάποιες καινοτομίες υπήρχαν αντιδράσεις. Πιστεύω βαθύτατα στην ικανότητα καινοτομία των επιχειρήσεων. Μπορούμε λοιπόν να αναλάβουμε κινδύνους, να διορθώσουμε τα ασφάλματα που υπάρχουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ε, χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέτρα ε, σαν πιδάλιο που θα μας οδηγήσει στο μέλλον για να δώσουμε σε ολόκληρο τον κόσμο και στην παγκοσμιοποίηση ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο γερουσιαστής κύριος Αλτάβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα έναντι του συναδέλφου από τη Ρουμανία που μίλησε για το γεγονός ότι σε ορισμένε επιχειρήσεις οι Ρωμά δεν μπορούν να εργαστούν. Εμείς το απογορεύουμε μέσω συντάγματος, αλλά θα ήθελα να πω ότι οι Ρουμάνοι στην Ισπανία είναι πάρα πολλοί και έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως κάθε εργαζόμενος. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να λυθεί ένα τέτοιο πρόβλημα ζωτικής σημασίας. Η Ισπανία επέλεξε μία λύση, η οποία απορρέει από τη συνένεση. Δηλαδή υπάρχει πραγματική θέληση υλοποίησης από τα συνδικάτα, τις επιχειρήσεις, τον ακαδημαϊκό κόσμο και ούτω καθεξής. Θέλουμε λοιπόν να εφαρμόσουμε αυτό, αυτή τη διακήρυξη. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε όλη την ε, εργασιακή αλυσίδα. Η ισπανική κοινωνία είναι πολύ απαιτητική και είναι πολύ υπεύθυνη έναντι των επιχειρήσεών της. Άρα εφαρμόζεται η διακήρυξη και σε επίπεδο επιχειρήσεων και ορισμένες ε, ΜΜΕ εκτός από τη συμμόρφωση, εκτός από την compliance έχουν ε, εντάξει και την Παγκόσμια Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η κυρία Αλμπορνός. Ευχαριστώ. Όπως ξέρετε το Εκουαδόρ ε, έχει την ευθύνη διαπραγμάτευσης του νέου μέσου και βρίσκομαι σε πολύ προνομιακή θέση να συμμετέχω και εδώ μεταξύ σας αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να είναι πιο ε, συμμετοχικές, θα μπορούσα να πω, σε αυτό το δεσμευτικό μέσο. Γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου θα ήθελα να συμμετάσχετε ενεργά από όλα τα εθνικά κοινοβούλια, γιατί η συνένεση είναι ύψης της σημασίας για την ε, εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη της να συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση αυτού του υποχρεωτικού μέσου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις συνεισφορές σας. Ευχαριστώ όλους τους βουλευτές, κυρίους και κυρίες. Νομίζω ότι ήταν καλή αυτή η συζήτηση. επ' τη ευκαιρία του ορτασμού της διακηρύξεως ε, της συνθήκης των, του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεός μαζί σας. Eh, Πάμε στο επόμενο πάνελ. Βιώσιμη ανάπτυξη και ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε τη χαρά και τιμή να έχουμε μαζί μας τον Ai Weiwei. Τον καλέσαμε να μας μιλήσει για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως είδαμε το πρωί, πολιτικοί φορείς και εκπρόσωποι συμφερόντων εξέφρασαν απόψεις στα πνεύματα της, στο πνεύμα της ε, διακήρυξης οικουμενικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται περί πολύ σημαντική συνιστόσα τη δημοκρατική κοινωνία θεμελιώδη είναι και η ελευθερία τη έκφραση, ο λόγο, η σημασία που έχει ο πολιτισμό στη δημοκρατία. Και γι' αυτό είναι προνόμιο για μένα να δώσω το λόγο σε ένα φιλοξενούμενο τόσο σημαντικό, όπως ξέρετε, ο Ai Weiwei είναι Κινέζος καλλιτέχνης που ασχολείται με τη γλυπτική ε, θές φωτογραφία, κινηματογράφο, κοινωνική κριτική, πολιτική κριτική, πολιτιστική κριτική μέσω των έργων του συμβάλλει συνεχώς στη συζήτηση τη δημόσια και την υποστήριξη αυτής της δημόσιας συζήτησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τη δημοκρατία. Τον ευχαριστώ που δέχτηκε να συμμετάσχει στο διάλογό μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του δίνω το λόγο αμέσως. Έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, στον πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκεται το ερώτημα του τι σημαίνει το να είναι κανείς άνθρωπος το να είμαστε άνθρωποι έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Η ανθρώπινη αυτοεπίγνωση και οι πράξεις για να σεβαστούμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι αυτό που δείχνει ιδιαίτερο νόημα στην ανθρωπιά. Η αυτοεπίγνωση και οι ανθρώπινες πράξεις ε, ε, εντάσσονται στην ε, αλληλεπίδραση μεταξύ ατομικής σκέψης και γλώσσας και της κοινωνίας εν γέννη βρίσκονται στα θέματα της οικονομικής ασφάλειας, στο δικαίωμα της, στην εκπαίδευση, στο δικαίωμα του συνεταιρίζεστε και στην ελεύθερη έκφραση. Οι ανθρώπινες πράξεις δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να προστατεύσουμε την ελεύθερη έκφραση και να ενθαρρύνουμε την θαραλέα σκέψη. Αν εγκαταλείψουμε τις προσπάθειες για το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, παρετούμεθα από το βασικό νόημα του να είμαστε άνθρωποι. Και όταν παρετούμεθα από τη δέσμευσή μας για την ιδέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκαταλείπουμε τις ηθικές από μια τέτοια αποτυχία προκύπτει διπροσωπεία και απερισκευσία, ε, διαφθορά και τυραννία και ανθρωπιστικέ κρίσει, όπω αυτέ, που αντιμετωπίζουμε στον κόσμο σήμερα. Έχουν περάσει πάνω από δύο αιώνε από τότε που προτάθηκε για πρώτη φορά η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτή την περίοδο η ανθρωπότητα έχει περάσει από διάφορα στάδια ιστορική ανάπτυξη και έχουμε δει τεράστιε αλλαγέ. Στην Ευρώπη που αρχικά είχαμε διάφορα απεικιοκρατικά και απολυταρχικά καθεστώτα. Έχουμε τώρα μια δημοκρατική κοινωνία με καπιταλιστικό προσανατολισμό που δημιουργεί ένα δημοκρατικό πλαίσιο και ένα μηχανισμό που προστατεύει τα ατομικά δικαιώματα. Μέσα στη νέα τάξη της παγκοσμιοποίησης ε, υπάρχουν διαρθρωτικές αλλαγές και η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Οι προκλήσεις ξεκινάνε από διάφορα αιτήματα κρατών σε διάφορα στάδια ανάπτυξης με διαφορετικές οικονομικές ε, καταστάσεις και ανταγωνιστικά οικονομικά συμφέροντα. Αλλά προκύπτουν επίσης προκλήσεις από διαφορετικές ε, αντιλήψεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, διαφορετικές αντιλήψεις για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα χρηστά και την υπευθυνότητα και διαφορετικέ ερμηνείε και εφαρμογέ των βασικών αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο σύγχρονο κόσμο, όσο αποδυναμώνεται ε, η φροντίδα μα για τι θεμελιώδει αξίε των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διακινδυνεύουμε να χάσουμε την ε, δυνατότητά μας να σεβαστούμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ιστορία μας δείχνει ότι μια τέτοια ηθική αποτυχία πάντοτε συνοδεύεται από επώδυνη πραγματικότητα. Η προσφυγική κρίση επιδεινώνεται καθημερινά και 70 εκατομμύρια πρόσφυγες αναγκάστηκαν να φύγουν από την κατοικία τους λόγω πολέμων και φτώχειας. Το ε, περιβάλλον μας ε, συνεχώς υποβαθμίζεται και η οικολογική ισορροπία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη. Ένοπλε σειράξει ε, παραμένουν, πολιτικές κρίσεις ελοχεύουν, περιφερειακέ ανισότητε, περιφερειακή αστάθεια οξύνονται. Αυτοκρατικά, αυταρχικά καθεστώτα ναι. επιβάλλουν με βία την θέλησή τους, ενώ η δημοκρατική διακυβέρνηση ε, παρακμάζει. Η ανετιολόγητη και ασίδωτη ανάπτυξη κάτω από την εθνικιστική και καπιταλιστική τάξη οξύνει το χάσμα μεταξύ φτωχών και πλουσίων. η εικόνα μας για τον κόσμο είναι διηρημένη και έχουμε όλο και περισσότερες διενέξεις από ό,τι στο παρελθόν. Σε πολλές χώρες και περιφέρειες του κόσμου δεν υπάρχει καμία ευκαιρία για τους ανθρώπους να έχουν παιδεία, δεν έχουν ευκαιρία να έχουν πρόσβαση στις ε, πληροφορίες ή στην επικοινωνία, ούτε να ασκήσουν την φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους και να εκπληρώσουν προσωπικά και κοινωνικά ιδεώδη. Δεν έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν η ελευθερία πεπιθήσεων και ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Τέτοια δικαιώματα και ελευθερίες αποτελούν ε, μια ε, θανάσιμη απειλή για τα απολυταρχικά καθεστώτα ε, και τον αυταρχισμό. Και γι' αυτό σε τόσο πολλούς χώρους φυλακίζονται οι δικηγόροι, εξαφανίζονται δημοσιογράφοι, δολοφονούνται δημοσιογράφοι η λογοκρισία έχει γίνει διαβρωτική, θρησκευτικές και μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, καταπιέζονται και διαφερμένα καθεστώτα συνεχίζουν να υποφελούνται από επισφαλείς ε, συνθήκες ε, με απερίσκεπτες πωλήσει όπλων και οι δικτατορίες έχουν την υποστήριξη των καπιταλιστικών εθνών οι θρησκευτικέ διαφορέ, ε, οι εθνοτικέ αντιφάσει και οι περιφερειακέ ε, διαφορέ ε, τροφοδοτούν αυτού του πρωτόγονου συσχετισμού ισχύω. Και η λογική είναι απλή. Όταν αποδυναμώνονται οι προσωπικέ ελευθερίε και εντείνονται οι έλεγχοι από τι κυβερνήσει, εντείνονται οι έλεγχοι από τι κυβερνήσει και τι κυριαρχούσε ελίτ. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι οι άνθρωποι δεν έχουν πλέον το δικαίωμα στη ζωή, δεν έχουν βασικέ ελευθερίε δεν είναι ελεύθεροι από φόβο, δεν έχουν την ελευθερία τη έκφραση, ούτε έχουν το δικαίωμα να έχουν ένα ελάχιστο πλαίσιο διαβίωση. Η έννοια των ανθρώπινων δικαιωμάτων πρέπει να αναθεωρηθεί. Οι συζητήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα επικεντρώνονταν στην μονοδιάστατη σχέση μεταξύ ε, των δικαιωμάτων του κράτου και των δικαιωμάτων του πολίτη. Αλλά τώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν μια πολυδιάστατη ε, σχέση και πολλέ επιπτώσει. Ανεξάρτητα ανεξάρτητα από το πώς εκφράζονται τα, δικαιώματα, όλα τα θεματολόγια βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και σε σχέση με άλλες περιόδους στην ιστορία μας οι συνθήκες που διέπουν την ανθρώπινη ύπαρξη ε, έχουν μεγαλύτερη διασύνδεση μεταξύ τους παγκοσμίω. Το δικαίωμα των παιδιών να μεγαλώνουν και να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Το δικαίωμα των γυναικών να είναι προστατευμένες. Το δικαίωμα της διατήρησης ε, του φυσικού περιβάλλοντος. Όλα αυτά είναι δικαιώματα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, άρρηκτα συνδεδεμένα με την επιβίωση του ανθρωπίνου είδους. Όσο εξελίσσονται η επιστήμη και η τεχνολογία, τα αυταρχικά κράτη εισβάλλουν ε, στον ιδιωτικό χώρο και περιορίζουν τις προσωπικές ελευθερίες στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της διατήρησης της σταθερότητας με ψυχολογική χειραγώγηση σε κάθε επίπεδο μέσω του ελέγχου του διαδικτύου και των ε, όλο και μεγαλύτερο έλεγχο και τελειοποίηση τη τεχνολογία της αναγνώριση προσώπου, τα αυταρχικά καθεστώτα εντείνουν τον έλεγχό τους ε, στη σκέψη και στις πράξεις των ανθρώπων και απειλούν ακόμη και με ε, εξάλληψη των πολιτικών δικαιωμάτων ομάδων οι οποίες επιζητούν την ελευθερία. Παρόμοια είδη ελέγχων επιβάλλονται ε, παγκοσμίω σε διαφορετικέ κλίμακε. Βλέπουμε ότι Υπό αυτές τις συνθήκες τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ε, είναι αντικείμενο μιας κοινή κατανόησης ε, ε, και δεν πρέπει η συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι στενή και κοντόφθαλμη. Σήμερα η Ευρώπη, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ρωσία, η Κίνα και άλλες κυβερνήσεις κατασκευάζουν έχουν στην ιδιοκτησία τους και πολλούν ε, όπλα. Εάν δεν καταφέρουμε να μειώσουμε αυτές τις επικίνδυνες πρακτικές ε, που κάνουν τις ένοπλες σειράξεις σε ολόκληρο τον κόσμο όλο και περισσότερο πιθανές ε, και εάν ε, δογματίζουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα απλώς, ε, οδηγούμαστε σε αυταπάτες. Αν δεν, υπάρχουν, αν δεν τεθούν όρια στην παγκόσμια εξάπλωση του καπιταλισμού και στη διαβρωτική διείσδυση της δύναμης του κεφαλαίου, αν δεν υπάρχει προσπάθεια να μειώσουμε την προσπάθεια των αυταρχικών κυβερνήσεων να ε, καταπολεμήσουν τις παρορμήσεις των ανθρώπων, οποιαδήποτε συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι κενά λόγια. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κοινέ αξίε, ανήκουν σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και εφόσον τα ανθρώπινα δικαιώματα ανήκουν σε όλου μα, όταν ε, παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, αυτό φύγει ε, ολόκληρη την ανθρωπότητα. Κατά αναλογία, μόνο όταν τα δικαιώματα όλων των ατόμων ε, σε ολόκληρη την ανθρωπότητα ε, είναι αντικείμενο μέρημνας και προστασίας, τότε η ανθρωπότητα μπορεί να οδηγηθεί σε μία λύτρωση. Αυτά είναι περί των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, που είναι μια απλή αρχή θα πρέπει να φτάσουμε σε μία συνένεση. Μήπως είμαστε πολύ βυθισμένοι στο, σκό, σκότος ή είμαστε πολύ εγωιστές ή δεν έχουμε το θάρρος. Μήπως ε, δεν είμαστε ειλικρινείς, ε, μήπως ε, γιατί δεν αγαπάμε τη ζωή αρκετά. Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και φανταζόμαστε ότι μπορούμε να ξεφύγουμε χωρίς να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας για τη δικαιοσύνη και την ευθυκρισία. Κοροϊδευόμαστε πιστεύοντας ότι μπορεί και να είναι αποδεκτό το χάος και δεν βλέπουμε ότι αυτό ε, καταστρέφει τα όνειρα και τις ελπίδες. Εάν πιστεύουμε πραγματικά στην ύπαρξη των αξιών και αν ε, ε, αναγνωρίζουμε την αλήθεια, αν κατανοούμε την επιστήμη, τον, το κάθε άτομο, αν υπάρχει σεβασμός για τη ζωή και επίσης την κοινωνία, τότε θα πρέπει να καταπολεμήσουμε κάθε εμπόδιο σε ένα θεμελιώδη ορισμό της ανθρωπότητας και θα πρέπει να τονίσουμε τις κοινέ μας αξίες για την ανθρώπινη ζωή, τη ζωή και του ανθρώπου και άλλων όντων που ζουν σε μια συμβιωτική αλληλεξάρτηση με το περιβάλλον. Αυτή, αυτό είναι το θεμέλιο για όλες τις ανθρώπινες αξίες και όλες τις ανθρώπινες προσπάθειες. Ευχαριστώ. Grazie. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να δώσουμε το λόγο στους βουλευτές. Συνάδελφε Μπέντλο από τη Ρουμανία. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε όλοι εδώ. Ευχαριστούμε για τις συνεισφορές που ακούγονται. Όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα είναι σημαντικό να κρατάσουμε εκ του σύνεγγυς τα πολιτιστικά δικαιώματα που είναι συνιστόσα σημαντική των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κοινότητε που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά τη διαμόρφωση πολιτικής που έχει σαν στόχο τα γλωσσικά δικαιώματα, πολιτιστικά δικαιώματα. Και η κοινότητά μα είναι τέτοια στη Ρουμανία. Εξακολουθούμε να επικαιροποιούμε την εθνική νομοθεσία, τόσο ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη τι πολιτιστικέ ανάγκε που έχουμε όσον αφορά την παιδεία και τη χρήση των μητρικών γλωσσών στα διάφορες περιοχές ε, των μειονοτήτων. Είναι κοινό τόπος ότι όλα είναι αλληλένδετα και η άνεση μιας κοινότητας επηρεάζει την περιφερειακή ανάπτυξη και συμβάλλει αυτή στη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει πολλαπλότητα προσεγγίσεων όσον αφορά τον πολιτισμό, τη γλώσσα και τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπάρχουν μεγάλες διαφορές ε, μεταξύ διαφόρων κοινοτήτων και πιστεύουμε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική απαιτείται που θα, θα είναι πιο φιλική για τις μειονότητες και αντικατοπτρίζει καλύτερη την πραγματικότητα για τις κοινότητες. Οι προκλήσεις της σύγχρονης εποχής ε, βάζει νέες, ε, νέα προβλήματα για τις κοινότητες στην Ευρώπη, οπότε χρειάζονται νέα ευρωπαϊκά πρότυπα για τις μειονότητες. Και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει στο μέλλον να εξετάσει τα πρότυπα αυτά για να προστατεύεται η ποικιλότητα που παρέχουν οι εθνικές μειονότητες στην Ήπειρο. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Άντζελα Γκουέρα. Καλημέρα σας και ευχαριστώ Ήθελα να συγχαρώ τον Ai Weiwei για την εξαιρετική του εργασία και θα ήθελα να πω ότι η Ατζέντα 2030 επιβάλλει στις χώρες να εφαρμόσουν και να τηρήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Πορτογαλία. Αυτό ακριβώς ε, γίνεται ή προσπαθούμε να το κάνουμε και μέσα στα πλαίσια της διμερού συνεργασίας τον, ε, ε, με τις χώρες που μιλούν την πορτογαλική γλώσσα. Ο τομέας της υγείας ε, μας απασχολεί ιδιαίτερα. Είναι επιτακτική η ανάγκη μέσα στα πλαίσια της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Εγώ συμμετείχα σε ένα τέτοιο φόρουμ στο Κιγκαλί, στη Ρουάντα. Βλέπω ότι οι αξίες είναι διαφορετικές στους μεν και στους δε, αλλά μία από τις ε, μεγαλύτερες δυσκολίες ε, για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η πρόσβαση στις βασικές ε, υπηρεσίες υγείας αλλά και αναπαραγωγής μέσα στα πλαίσια του δημογραφικού που απασχολεί την Ευρώπη. Άρα θα θέλαμε να δούμε ποια ε, χρηματοδοτικά μέσα υπάρχουν από τα Υπουργεία σε εθνικό επίπεδο και θεωρώ ότι δυστυχώς υπάρχουν πολλές περίκοπες κονδυλίων στον τομέα της υγείας και θα ήθελα να πω πώς προωθείτε την εγγύηση αυτών των δικαιωμάτων ε, μέσα στα πλαίσια των στενοπών που έχουν δημιουργηθεί. Επίσης, η ατζέντα των ε, μεταναστευτικών ροών επιβάλλει αυτό ως πρωταρχικό μέλημα την πρόσβαση στον τομέα της υγείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αρκεστείτε στο ένα λεπτό. Μπάρμπαρα, δώσε το σωστό παράδειγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δήλωσή σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω που χρησιμοποιείτε την τέχνη σας και την πολιτική σας σκέψη και αντίληψη για να μπορείτε να κρίνετε και να επικρίνετε και να προσπαθείτε να βελτιώσετε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κλειστά σύνορα. Εμείς τα κράτη-μέλη και διάφορες οργανώσεις έχουμε αποτύχει κτρά στο να εφαρμόσουμε το δικαίωμα της προστασίας για τους πρόσφυγες στα σύνορά μας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα ευρωπαϊκά σύνορα είναι τα πιο θανατηφόρα στον κόσμο. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ. Δεύτερον, αναφερθήκατε σε μια έννοια. Την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει κανείς να είναι ελεύθερος από το φόβο, είπατε. Το φόβο της κυβερνήσεως, αλλά και φτωχό δεν πρέπει να είσαι ελεύθερος από τη φτώχεια. Και αυτή είναι η ουσία όταν συνετάχθη η διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα βλέποντας την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και την πρόσφατη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτή η αντίληψη αντικατοπτρίζεται, πιστεύω. Δεν χρειάζεται μια νέα σύνταξη κειμένου, πρέπει η ιδέα να εφαρμοστεί σωστά. Και αν δείτε το σχέδιο δράσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα το δείτε ότι χρειαζόμαστε και τα δύο. Δεν μπορεί να ζήσει κανείς μια αξιοπρεπή ζωή χωρίς να είναι ελεύθερος από τη φτώχεια και να είναι ελεύθερος από το φόβο. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει καλή δουλειά. Προωθεί αυτό, αυτή την έννοια, αλλά καμιά φορά βέβαια πέφτουμε στη ρητορική ξανά του ψυχρού πολέμου και πιστεύουμε ότι τα πολιτικά δικαιώματα ε, είναι πιο σημαντικά από τα άλλα και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει σε διεθνές επίπεδο όπως το νοεί της προσπάθειας. ούτως ώστε η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να προωθείται όταν τα ατομικά και τα συλλογικά δικαιώματα είναι εγγυημένα μαζί, μόνο τότε. Με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σουσκίν, συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς και εγώ να ευχαριστήσω τον Ai Weiwei, όπως και άλλοι που είναι μαζί μας σήμερα, που ήρθε να μιλήσει στο Ευρωκοινοβούλιο και δεν μπορεί να μιλήσει και να εκφραστεί στη χώρα του. Ήδη αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό σημάδι που δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει αυτό το μήνυμα για τη σημασία και το ρόλο που παίζουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά το θέμα αυτό. Αναφερθήκαμε στο βραβείο Ζαχάροφ ε, που οδήγησε σε απονομή βραβείο Νόμπελ ε, Ειρήνης. Είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτός ο διάλογος μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Δεν μπορούμε παρά να ανταλλάσσουμε εμπειρίες έτσι. Να σας πω δύο πρωτοβουλίες που αναφέρω που έχει αναλάβει το κοινοβούλιο μας στο Βέλγιο. Μια πρωτοβουλία, ένα μικρό το γαλλόφωνο Βρυξε... Ε, κοινοβούλιο των Βρυξελών υιοθέτησε ένα ψήφισμα που στηρίζει τη διευκόλυνση ω ανθρωπιστικής θεώρηση διαβατηρίων, βίζας και να μην ποινικοποιείται η αλληλεγγύη που παρουσιάζουν οι πολίτες στους πρόσφυγες και αλληλέγγυα πολιτική μετανάστευση και βιώσιμη σε ένα πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε τη Σύνοδο Κορυφή για τη μετανάστευση στο Μαρακέ και δήλωσαν πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε ότι θα αρνούσαν να υπογράψουν το σύμφωνο αυτό, που δεν είναι ένα σύμφωνο υποχρεωτικό στην εφαρμογή του. Και στο Βέλγιο γίνεται συζήτηση μεταξύ κάποιων κομμάτων της πλειοψηφία και του Πρωθυπουργού και Εθνικιστικού Κόμματο που αρνούνται το Βέλγιο να υπογράψει, ενώ ο Πρωθυπουργό είχε δεσμευτεί είναι ανοιχτή η εκκρεμή συζήτηση. Δράτω με τι ευκαιρίε τη συναντήσεω για να ενημερώσω του συναδέλφου ότι διοργανώνουμε εδώ στι Βρυξέλλε σε, ε, σε διάφορα βήματα ένα συμπόσιο σημαντικό για την κατάσταση στον Μπουρούντι. Διότι είναι ένα από τα παραδείγματα όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα προφανώ δεν γίνονται σεβαστά, διότι ο πρόεδρο αρνήθηκε να τηρήσει υποχρεώσει ενώ έχει υπογράψει στην ε, αρούσα μια δέσμευση να μην είναι υποψήφιος για δεύτερη θητεία και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες του Μπουρούντι τώρα είναι πρόσφυγες σε γειτονικέ χώρες και στη διασπορά και εδώ στις Βρυξέλλες θα έχουμε πάνω από 80 ε, κατοίκους του Μπουρούντι που είναι από καταβλισμούς ε, προσφύγων έρχονται από τον Μπουρούντι και από την Ευρώπη να συζητήσουν την κατάσταση και κυρίως την έρευνα που ξεκίνησε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο όσον αφορά την κατάσταση του Μπουρούντι μία μέρα πριν το Μπουρούντι αποχωρήσει από το δικαστήριο. Όσοι ενδιαφέρονται από τους συναδέλφους, ε, σας λέω ότι υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία και σας ενημερώνω και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Συνάδελφε Κάνουν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Άι Βεβέι, είναι χαρά. Μου πολύ όμορφα σέλφις έχετε εμπνεύσει κόσμο στον κόσμο, με τη... όλο τον κόσμο, στην Ιφίλιο, με την τέχνη σας. Ζωγραφίζετε ειλικρινή εικόνα για την κατάσταση στον κόσμο, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για τις μειονότητες στην Κίνα, τους Τιβετιανούς και αυτά που συμβαίνουν με τις μειονότητες. Μέσω τέχνης μπορείτε να εμπνεύσετε τον κόσμο Όμως οι πολιτικοί λαμβάνουν αποφάσεις για μια χώρα. Τα κινήματα είναι υπέροχα, λαμπρή τέχνη, πολύ ισχυρή. Αλλά πώς μπορείτε να μεταφράσετε εσείς το έργο σας που εμπνέει, ούτως ώστε να αλλάξουν απόψεις στα κοινοβούλια στον κόσμο εκεί σε χώρες που υπάρχουν προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι μπορείτε να κάνετε, σε ποιο βαθμό μπορείτε να κινηθείτε, να προσπαθήσετε σε ποιο βαθμό εργάζεστε στο επίπεδο των κοινοβουλίων και των πολιτικών για να του επηρεάσετε. Σταματάκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κυρίες και κύριοι, ε, στο πλαίσιο της Ειδικής Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο του 2015 υιοθετήθηκε από τους αρχηγούς κρατών η Ατζέντα 2030 με τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Η επίτευξη αυτών των στόχων απαιτεί μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης και παγκόσμια συνεργασία ώστε να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό οι τρεις άξονες ανάπτυξης, ο οικονομικός, ο περιβαλλοντικός και ο οικονομικός. Στα πλαίσια αυτά και μέσα στο λίγο χρόνο που έχω ε, θέλω να σας παρουσιάσω ε, κάποιες πρωτοβουλίες που έχουν επαρθεί από τη χώρα μου, από την Ελλάδα. Το Υπουργείο Παιδείας δραστηριοποιείται στους τομείς ειρήνης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανάπτυξης, της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, της παγκόσμιας ηθαγένειας και της παγκόσμιας κληρονομιάς. Στην Ελλάδα πρόκειται να υιοθετηθεί ένα νέο σχέδιο δράσης για το παιδί, το οποίο όχι μόνο θα συμβάλλει στην καλύτερη προστασία αυτής της ευάλωτης ομάδας, αλλά και γιατί για πρώτη φορά το παιδί αντιμετωπίζεται ως ένας νεαρός πολίτης και όχι ως παρακολούθημα το γονιό του. Στο επόμενο στάδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρόκειται να δοθεί έμφαση στην αρχή της ίσης μεταχείρισης που συνδέεται άμεσα με την αντιμετώπιση της φτώχειας την ελεύθερη πρόσβαση σε ισότιμη εκπαίδευση, την ισότητα των φύλων, την εξάλληψη των ανισοτήτων, τη δημιουργία βιώσιμων και δημοκρατικών πόλων και την ανάπτυξη μιας δίκαιης κοινωνίας. Πολύ σημαντικό βήμα για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα πλαίσια του μοντέλου ανάπτυξης όπως το περιγράψαμε ε, είναι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού της χώρας μας ε, για την εγγραφή στο Μητρό Ανέργων ομάδων ανέργων που στενούνται μόνιμης κατοικία ή διαμονής. Με αυτή την απόφαση οι άνεργοι πρόσφυγες που ζουν σε διάφορες δομές προσωρινές φιλοξενίας. Οι άνεργοι άστεγοι, οι άνεργες γυναίκες που φιλοξενούνται σε ξενώνες είναι θύματα ε, ε, βίας ενάντια στις γυναίκες. Οι άνεργοι ζέοι, νέοι που ζουν σε δομές παιδικής προστασίας ε, και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν σπουδάζουν και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία είναι άνεργοι και φιλοξενούνται σε μονάδες ψυχικής υγείας και αποκατάστασης έχουν τη δικαιότητα τη δυνατότητα να εγγραφούν στο Μητρό και να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την ομιλία σας που είναι πηγή έμπνευση. Πιστεύω ότι καλά κάνουμε και αναφερόμαστε στην τέχνη, γιατί δεν, δεν δίνουμε αρκετή σημασία στο ρόλο που παίζει η τέχνη, η λογοτεχνία ή οποιαδήποτε άλλη μορφή τέχνης. Αναφέρθηκα στην ασυνέπεια της πολιτικής μας προηγουμένως. Χρησιμοποίησαμε το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σημαντικός δωρητής βοήθειας και ταυτόχρονα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν στο εμπόριο όπλων. Δεν δόθηκε καμία απάντηση όταν το έθιξα εγώ στην προηγούμενη ομιλία μου, στην προηγούμενη συνεδρία. Χαίρομαι λοιπόν που το αναφέρετε εσείς στην ομιλία σας στο θέμα του εμπορίου όπλων. όταν βλέπουμε την αντιμετώπιση της μετανάστευσης ε, και ε, το θέμα των κέντρων κράτησης ε, στη Λιβύη, όπου υπάρχει κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλα αυτά πρέπει να τα στυλιτεύσουμε. Αναφέρθηκαν οι στόχοι τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπου περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση. Πρέπει να είναι ποιοτική εκπαίδευση. Δεν θέλουμε απλώς μεγάλο αριθμό παιδιών στα σχολεία, θέλουμε να παίρνουν και ποιοτική εκπαίδευση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Αϊβαϊβέη, ε, να σας ευχαριστήσω για την ε, ε, δράση σας παγκοσμίω σε θέματα οικολογίας και διατήρησης ενός σωστού χώρου διαβίωσης για τους ανθρώπους. Έχω ε, την εξή ερώτηση. Τι συμβολή μπορεί να έχει η τέχνη, πώς μπορούν να συμβάλλουν οι καλλιτέχνες για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την περαιτέρω ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Μιλήσατε για απειλές ε, στον ιδιωτικό χώρο των ανθρώπων ε, μέσω των ψηφιακών μέσων τεχνολογίας. Τι μέτρα μπορεί να λάβει η πολιτική για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σέγκελ, Μια παρόμοια ερώτηση έχω κι εγώ. Οι καλλιτέχνες, ε, οι σκηνοθέτες, ε, πολύ συχνά στο πλαίσιο ανοιχτών συζητήσεων ε, αναφέρουν πολλά άλλα και όχι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι λίγοι οι καλλιτέχνε ε, που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διάσημοι καλλιτέχνε όπω ο Damian Hirst, παραδείγματο χάρη, δεν άκουσα ποτέ να μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά τη γνώμη σα, γιατί οι καλλιτέχνε δεν μιλάνε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 7-8 λεπτά για να απαντήσετε. Ε, άκουσα αυτά που υπόθηκαν. Άκουσα να αναφέρονται τα δικαιώματα των παιδιών, τα δικαιώματα των γυναικών, των μειονοτήτων παιδιών. Αυτές οι συνιστώσεις της κοινωνίας είναι ένα κομμάτι του μέλλοντος. Χωρίς τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών, των μειονοτήτων, όπως είναι οι Θιβετιανοί και η Βίγκα και η προστασία των δικών τους δικαιωμάτων, τότε η συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ατελής και δεν μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας. Ε, βέβαια, μέσω νομοθεσίας και σε δικαστικό επίπεδο και σε επίπεδο διαμόρφωσης πολιτικής και κυβερνητικό επίπεδο πρέπει όλοι αυτοί οι τομείς να βελτιώσουν το έργο τους και να αλλάξουν. Πολλές κυβερνητικές αλλαγές προέρχονται από πιέσεις που ασκούν άλλες κυβερνήσεις. Και αυτή η πίεση μπορεί να είναι διαφόρων ειδών, μπορεί να είναι οικονομική πίεση, μπορεί να είναι άλλα είδη πίεσεως. Και μέσω των φωνών και των πιέσεων θα αλλάξουν οι χώρες. Πολύ σπάνια αυτές οι αλλαγές συνέβησαν με φυσικό τρόπο. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω γιατί η τέχνη είναι ένας ενδεχόμενος τομέας για την προώθηση ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι όταν ζει κανείς σε μια φτωχή κοινωνία, τότε τα αισθήματα του κόσμου επικρατούν. Θέλει ο ένας να συμπεριφέρεται σωστά στον άλλον. Αυτό είναι είναι κοινό για όλους. Το βλέπει κανείς σε όλες τις κοινωνίες. Δηλαδή ότι ε, μόνο η τέχνη μπορεί να βρει αυτό τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Στην πολιτική, την οικονομική σφαίρα υπάρχουν πολλοί λόγοι που οδηγούν στο να αγνοεί κανείς το πιο βασικό, το πιο σημαντικό ε, όρο για την ανθρώπινη ζωή. Τη δυνατότητα να αισθάνεται κανείς και να συλλαμβάνει αισθητικά μηνύματα. Ε, και αυτά, αυτά τα συναισθήματα και οι αισθήσει ε, έχουν σχέση ε, με τα συναισθήματά μας. Η τέχνη μπορεί να βρει τον άνθρωπο να καταλάβει τις πιο βασικές αλήθειες. Και η τέχνη μπορεί να επιτρέψει να βρούμε και να διερευνήσουμε δυνατότητες. Να ανακαλύψουμε τα εσωτερά μας αισθήματα τα συναισθήματά μας τα ενδόμηχα. Ε, και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει η πολιτική. Υπάρχουν, γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί καλλιτέχνες που δεν μιλάνε για τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν ένα άλλο ερώτημα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό. Ένας λόγος είναι η παιδεία. η παιδεία πολύ συχνά διαχωρίζει την πολιτική από την τέχνη, από άλλους τομείς. Ε, φοβούνται ίσως ότι η πολιτική είναι ασύμβατη με την τέχνη. Ή ότι η πολιτική σχετίζεται με τη διαφθορά, ότι, η πολιτική είναι κάτι λάθος. Αλλά ο πολιτισμός, η κουλτούρα και η πολιτική είναι πάντα ε, αλληλένδετα. Οι καλύτεροι λοιπόν θα πρέπει να εστιάζονται επικοινωνικών ζητημάτων και επί της καταστάσεως για τους ε, λαούς κάθε κοινωνίας και να συγκεντρώνονται και στα συναισθήματα των ανθρώπων αυτών. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε εδώ με αυτά τα λόγια, πάρα πολύ σημαντικά λόγια που εξέφρασε ο κ. Ευχαριστώ όλους τους φιλοξενούμενους μας, τους συμμετέχοντες της ομάδας εργασίας που είναι εδώ μαζί μας σήμερα, που μοιραστήκανε μαζί μας την εμπειρία τους, τις σκέψεις τους. Ήταν η ιδιαίτερη μέρα για όλους μας, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Η δουλειά που έγινε από τις τρεις ομάδες ενώθηκαν από ε, ε, έναν μύτο της Αριάδνης που έδειξε πώς μπορούν να κινηθούν τα εθνικά κοινοβούλια συνεργασία με το Δημόσιο Κοινοβούλιο και τι προσπάθειες μπορούν να καταβληθούν για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του ατόμου και κυρίως στα πλαίσια της εξωτερικής ε, πολιτικής πρέπει να παγιώνονται αυτές οι αρχές και συνεχώ μπορούμε να τα προωθούμε και να είμαστε περήφανοι για τι αρχέ. Ευχαριστώ πραγματικά του επιφανεί ομιλητέ και όλου του φιλοξενούμενου που συμμετείχαν στη συζήτηση σήμερα το πρωί. Θέλω να καλέσω όλου να συμμετάσχετε στην εκδήλωση υψηλού επίπεδου που διοργανώνεται από την ευκαιρία τη 70η επαιτίου τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ξεκινήσει το απόγευμα στι 2.30 στην αίθουσα τη Ολομέλεια, στο ημικύκλιο εδώ. Και κάτι οργανωτικό ίσως προσκεκλημένους για το γεύμα, θα πρέπει να πάτε στο εστιατόριο των Ευρωβουλευτών. Σας ευχαριστώ εκ νέου για τη σημαντική μέρα, το σημαντικό πρωινό. Καλή συνέχεια εύχομαι σε όλους και καλή σας όρεξη.